ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα τον ε, Υπουργό Υπεύθυνο για Ευρωπαϊκά Θέματα, κύριο Διέγκο Λόπεθ Καρίγιο, από την Ισπανία βεβαίως, και γνωρίζουμε, τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι τον είδαμε στα πρώτα έδρανα της Ολομελίας του Στρασβούργου για πολύ σημαντικά θέματα πρόσφατα. Είναι εδώ λοιπόν μεταξύ μας ο κύριος Υπουργός έτσι ώστε να μας, αναπτύξει, να μας αναπτύξει συγγνώμη, το όραμά του, τις απόψεις του, ε, το πρόγραμμα εργασίας ε, επί του οποίου εργάζεται. Βεβαίως θα θέλαμε να κάνετε αναφορά και στην στρατηγική του 2020, γιατί τον Απρίλιο ξεκινάμε με μια σειρά σημαντικών διασκέψεων. Τον Απρίλιο θα ακολουθήσει άλλη τον Ιούλιο και για το θέμα αυτό ο κύριος Μόντι θα κάνει συγκεκριμένη έκθεση. Στις 7 ε, Απριλίου θα υπάρξει ειδική ολομέλεια του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να συζητήσουμε τα της διασκέψεως ε, κορυφής. Αυτά είναι καλά. Βέβαια το άσχημο είναι ότι οι εργασίες τη Επιτροπή μα θα γίνουν από τι 4.30 μέχρι τις 8 το βράδυ και αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο, εν πάση περιπτώσει. Με ιδιαίτερη χαρά δίνω τον λόγο στον ε, Υπουργό, κύριο Λόπε Καρίγιο. Και καλώς ορίσατε βέβαια, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ. Μέλη της Επιτροπής της Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Αυτό το εξάμεινο έχουμε λάβει την Προεδρία του Συμβουλίου. Και την Προεδρία του Συμβουλίου Ανταγωνισμού και Ανταγωνιστικότητας. Οπότε, αποτελεί τιμή για μένα να σας επισκέπτομαι σήμερα για πρώτη φορά, ώστε να σας παρουσιάσω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Προεδρίας μας για τον τομέα της ε, πολιτικής ιστορικής αγοράς από πλευρά τη ισπανική κυβέρνηση. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συγκυρία μια που πρόκειται να έχουμε μια νέα νομική βάση για το σύνολο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι πρόσφατη η αρχή της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όπως ξέρετε, ανέλαβαν καθήκοντα μόλις πριν από δύο μήνες πρώτης ενάρξη της Ισπανικής Προεδρίας, οπότε και εμείς Κατά αυτό το εξάμεινο θέλουμε να ξανακερδίσουμε το χαμένο χρόνο, Αυτό που χάθηκε. Και λόγω των θεσμικών λαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και λόγω της ε, καθυστέρησης της ε, ε, ε έναρξη τη θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που του γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Οπότε θα πρέπει και εγώ να αναγνωρίσω δημοσία το έργο το οποίο επιτέλεσε η Σουηδική Προεδρία, αλλά επίση και το έργο το οποίο η, η Τρόικα, Ισπανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, τώρα επιτελούμε με τρόπο αλληλέγγυο, με συνέπεια και συνεργασία. Και έχουμε από κοινού ένα 18 μήνο πρόγραμμα. Οπότε θεωρούμε ότι προλυάνουμε το δρόμο τόσο ώστε να συνεχιστεί εύρεθμα οι πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαν συνέπεια της ε, συνθήκης της Λισαβόνας να έχουμε τώρα ένα πιο ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει καινούργιε νομοθετικέ ε, αρμοδιότητε, καινούργιε πολιτικέ αρμοδιότητε και ελεγκτικέ επίση. Και για αυτό το λόγο εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, μια που έχω την ευκαιρία σήμερα να τα πούμε μαζί. Μια που είστε πάρα πολύ σημαντικό συνομιλητή του Συμβουλίου. Είναι κάτι το οποίο θα λάβει χώρα για πρώτη φορά, μια που είναι τώρα η πρώτη Προεδρία που ασκεί τις αρμοδιότητές της υπό την ε, συνθήκη της Λεσσαβόνας, την καινούργια. Τώρα. Θα διαρθρωθεί η ομιλία μου γύρω από δύο άξονες. Πρώτα-πρώτα. Θα μιλήσουμε για τα της εσωτερικής αγοράς. Γενικώς Τι είναι η ιστορική αγορά. Είναι ένα από τα κοσμήματα, από τα στολίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης υποτέλεσε μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση. Μια μεγάλη κατάκτηση για αυτό τον πρώτο μισό αιώνα της διαδρομής, της ζωής της. Επίσης, είπαμε ότι τώρα ξεκινά μια νέα φάση στην, στον βίο, στην διαδρομή της εσωτερικής αγοράς. Ε, είναι πιο ενδιαφέρον, πιο σημαντικό το τοπίο τώρα. Τόσο το μάλλον που είναι τόσο σημαντική η εσωτερική αγορά, οπότε προς τα εκεί θα κινηθώ στο πρώτο μισό της ομιλίας μου και στη συνέχεια πρόκειται να σας πω ποιες είναι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το σχέδιο οδηγία, ε, υποδιαμόρφωση, ό,τι τέλο πάντων έχουμε στην πολιτική μα ατζέντα, που βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται. Θα συνεργαστούμε και φυσικά η δική σας Επιτροπή και είμαστε οι δύο συνομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινώ τώρα με μια πρώτη σκέψη μου όσον αφορά το πώς θα τονώσουμε την εσωτερική αγορά. Και όπως προανέφερα βρισκόμαστε υπό μια συγκυρία οικονομικής κρίσης. Πάμε να δούμε πώς θα πετύχουμε μια οικονομική ανασυγκρότηση, να δούμε πώς δεν θα παροξενθεί η, κατάκτη, η κρίση αυτή που είναι από τη δεκαετία του 30 πιο σοβαρή που σοβεί και οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε, να θωρακίσουμε την εσωτερική αγορά. Πώς θα μπορέσουμε να δούμε τις καινούργιες διαστάσεις του πράγματος και θεωρούμε ότι στα πλαίσια αυτά είναι πάρα πολύ θετικό το ότι η εσωτερική αγορά προβάλλεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Μαρτίου που αφορά την στρατηγική με τον ορίζοντα του 2020 για ανάπτυξη και απασχόληση. Επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι η... έχει πολλές πλευρές η ιστορική αγορά και φαντάζομαι ότι οι κρατών και κυβερνήσεων στην ε, πρώτη επίσημη συνάντηση. Θα το αναγνωρίσουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά και στην τελευταία θα επιβεβαιωθεί αυτό τότε που στην τελευταία ε, συνάντηση της Προεδρίας μας πρόκειται να αρχίσει επίσημα αυτή η στρατηγική του 2020, αυτά να γνωρίσουν, ήθελα να πω, ότι η εσωτερική αγορά είναι κάτι πάρα πολύ βασικό σαν στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως σας είπα, πρόκειται για αυτό το έγγραφο της 3 Μαρτίου, όπου αναφέρεται ότι σαν εργαλείο μέσω πολιτικής που έχει η Ένωση στα χέρια της είναι η εσωτερική αγορά από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά είναι τα ευρωπαϊκά ταμεία. Τα διαρθωτικά ταμεία Αυτά είναι τα δύο μεγάλα μέσα πολιτικής, τα δύο, τα δύο όπλα, τα δύο εργαλεία που έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει βέβαια με τον πιο δόκιμο τρόπο και πιο πρόσφορο να τα χρησιμοποιήσει. Πρόκειται για κάποιες καινούργιε διαστάσει που έχουν προσδοθεί στην εσωτερική αγορά. Επίσης, έχουμε συναντηθεί και συζητήσει με τον ε, παλαιό επίτροπο, τον κύριο Μαρία Μόντι. την 1η Μαρτίου στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού και Ανταγωνιστικότητα. Είχαμε επίση και ένα άτυπο γεύμα εργασία, ε, Συμμετέσχουν όλοι οι Υπουργοί Αρμόδιοι για την Ιστορική Αγορά και παρεκάθισε και ο κύριος Μόντι, ο καθηγητής Μόντι και επίση είχαμε και τον Αντιπρόεδρο και τον κύριο Ταγιάννη της Επιτροπής και, αλλά και τον Επίτροπο Μπαρνία που έχει το χαρτοφυλάκι της Αγοράς. Οπότε και υπό την αιγύδα του πρόεδρου του κ. Μπαρόσου θα ετοιμαστεί ένα κείμενο όσον αφορά το μέλλον τη ε, ιστορική αγορά. Αυτό ήταν ο στόχο τη συνάντηση, πώ θα εκπονηθεί αυτό το ε, πόνημα. Και ε, οπότε είπαμε ακριβώ ποια είναι τα θέματα που, που έχει κολλήσει ελαφρώ η ευρωπαϊκή οικοδόμηση και επίση είδαμε ποιοι, ποιοι κλάδοι τη οικονομία έχουν περισσότερο πληγή από την χρηματοπιστωτική κρίση. Ο δε καθηγητή Μόντι μίλησε ε, για την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ κοινή γνώμη και εσωτερική αγορά, ε, γιατί αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι ένα φραγμό για τα νέα βήματα προ τα εμπρό. Όμω είναι και μια ευκαιρία τόσο ώστε να προχωρήσουμε προ ε, αναβάθμιση, προ πρόοδο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και τα εξήγησε καθόλου τον τρόπο ο κύριο Μόντι, πρώτα-πρώτα για, για το θέμα τη αναζωογόνηση τη εσωτερική αγορά, ούτω ώστε να μπορέσουμε την ισχύουσα νομοθεσία να την ενεργοποιήσουμε. Από την άλλη μεριά είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για περισσότερη ολοκλήρωση στους τομείς εκείνους όπου ακόμα δεν έχουν θεσπιστεί ε, νόμοι, κανόνες και νομοθεσία γενικότερα διότι θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Και μας είπε ποιοι είναι οι τομεί, ποιε είναι οι διαστάσει τη εσωτερική αγορά, όπω οι υπηρεσίε, όπω τα θέματα τη ψηφιακή τεχνολογία, ε, η, η ενέργεια, οι μεταφορέ, οι τηλεπικοινωνίε, αυτέ οι πτυχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μα είπε ότι είναι η υλική δομή ούτω ή τη εσωτερική αγορά. Δηλαδή δεν είναι το νομικό μέρο, αλλά είναι το υλικό, το πρακτικό, το χειροπιαστό μέρος όπου έχουμε ε, εκεί για το πρόβλημα, διότι κάποιες φορές υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη διασύνδεση ε, και στις μεταφορές και στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, μας είπε για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για την εξωτερική επιτυχία της ιστορικής αγοράς, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την φάση στην οποία βρίσκονται και βεβαίως ε, όλες αυτές τις σκέψεις τις ενέταξε και στην προσπάθεια που κάνουμε για το περιβάλλον και την ε, ε, αλλαγή του κλίματος εν ώψη της ε, συνάντησης του Συμβουλίου Πέμπτη και Παρασκευή της επόμενης εβδομάδα. Ο Μαριό Μόντι ξεκάθαρα διευκρίνησε ότι πρέπει η εσωτερική αγορά να έχει πιο θετική υποδοχή εκ μέρου πολιτών και επιχειρήσεων. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο πιο καινοτόμο να γίνει αυτή η προσέγγιση του κόσμου με την ιστορική αγορά. Οπότε οφείλω να σας πω ότι σε εκείνη τη συνάντηση που είχαμε με ευκαιρία του Συμβουλίου με τον Μάριο Μόντι και του υπουργού για νομισμό και αγωνιστικότητα όλοι συμφωνήσαν με το πώ τα βλέπει τα πράγματα ο Μάριο Μόντι. Και είπαν ότι συμμερίζονται την άποψή του τόσο ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε να δώσουμε ένα νέο δυναμισμό στην εσωτερική αγορά. Οπότε, αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσει μια τέτοια διαδρομή. Μια τέτοια διαδρομή η οποία να χαρακτηρίζεται από αυτή την τόνωση τη εσωτερική αγορά. Οπότε. Νέα όθηση. Άρα. Θα πρέπει να δοθεί στην εσωτερική αγορά και συμφώνησαν οι υπουργοί μαζί του. Υπάρχουν δε ορισμένοι κλάδοι τη οικονομίας που μπορούν να βοηθήσουν στην αυτή την αναθέρμανση τη ιστορικής αγορά, όπως είναι ο τομέας των υπηρεσιών ή ο τομέας της ψηφιακής τεχνολογίας ή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης έχουμε την υποδομή που είναι σαν σπαδελική στήλη της ιστορικής αγοράς. Υπήρξε ζωντανή, ζωηρή, μεστή αυτή η ο τομεας της ψηφιακης τεχνολογιας η του ηλεκτρονικου εμποριου Επίση εχουμε την υποδομη που ειναι σαν σποδελικη στηλη της ιστορικης αγορας υπηρξε ζωντανη ζωηρη μεστη αυτη η συζητηση και γι' αυτό το λόγο η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου πρότεινε και έγινε αποδεκτή η πρόταση από τους υπουργούς. Αυτό το ζήτημα της αναθέρμανσης της ιστορικής αγοράς να συμπεριληφθεί ο σημείο της μίσας διάταξης του Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαΐου. Και έτσι να γίνει μια πρώτη συζήτηση, να διατυπούν κάποιε πρώτες ιδέες και σκέψεις πάνω στην ε, έκθεση του Μάριο Μόντι. Και η έκθεση αυτή τελικά να υποβληθεί στον Πρόεδρο Μπαρόσα. Τώρα να πούμε κάποια άλλα θέματα που έχουν απασχολήσει το Συμβούλιο και που επίσης τώρα απασχολούν το Κοινοβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για κάποια νομοθετήματα τα οποία τώρα βρίσκονται στην ε, φάση της τελικής ευθείας για την ε, θέσπισή τους ή στην φάση της εφαρμογής, όπως σε αυτή την περίπτωση η οδηγία για τις υπηρεσίες. Πολύ σημαντική η πρωτοβουλία. Τις πιο σημαντικές που έχει ποτέ θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τις υπηρεσίες που όπως γνωρίζετε καλά είναι περίπου το 70% του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Αλλά και όσον αφορά τη δημιουργία της απασχόλησης, εκπροσωπούν το ίδιο ποσοστό. Άρα, ό,τι και να πούμε δεν είναι υπερβολικό για τις υπηρεσίες. Θα, θα πρέπει επομένω να δούμε στο πλαίσιο τη εσωτερική αγορά, τι μπορούν να κάνουν αυτέ οι υπηρεσίε, ο τομέα των υπηρεσιών, ούτω ώστε να αναθερμάνουν την, την απασχόληση, την εσωτερική αγορά, για να ε, ανταποκριθούν οι υπηρεσίε σε αυτό που θέλουμε να ε, είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οπότε και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ό,τι δυνατότητε προσφέρει αυτή η οδηγία για τι υπηρεσίε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ μια ει βάθο μεταρρύθμιση. Οπότε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις αρχές που από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε όσο γίνεται διαφάνεια, να έχουμε όσο γίνεται νομοθετικό ευμενές κλίμα για τους εμπλεκόμενους, τους φορείς, τα νομικά φυσικά πρόσωπα, όλους όσους ενέχονται σε αυτές τις ε, υπηρεσίες. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό η σχετική οδηγία να μεταφερθεί στο ιστορικό δίκαιο και επίσης αυτή η μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο να είναι η πιο ενδεδειγμένη. Το 31 Δεκάτου εξέπνευσε σχετική προθεσμία. Όμως δεν μπορούμε να το κρύψουμε ακόμη δεν έχει γίνει η αναδοχή αυτής της οδηγίας σε όλα τα στεργαδίκια των κρατών μελών. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να γίνει αυτή η μεταφορά στο στεργοδίκαιο και να γίνει με τον πιο ορθό τρόπο. Ήδη όπως ξέρετε ισχύει ε, μία μέθοδος ε, αξιολόγησης, ελέγχου το πώς γίνεται αυτή η μεταφορά όπως ξέρετε προβλέπεται από το 39 αυτής της οδηγίας, γίνεται κάτι σαν αμοιβαία αξιολόγηση. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, οπότε και με αυτόν τον τρόπο, στο επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα μπορέσουμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, ούτως το Συμβούλιο Τη 25 η και 26ης Μαΐου να είναι αποδοτικό. Και γι' αυτό και στη μέση διάταξη προβλέπει να ζητηθεί και αυτή η διαδικασία τη αμοιβή αξιολόγηση. Επίση, με τη βάση τη έκθεση τη Κομισιόν θα δούμε τι λέει η Κομισιόν για την μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο τη οδηγία για τι υπηρεσίε. Τώρα, να σα πω και αυτό το σχέδιο τη οδηγία όσον αφορά τη την υπερημερία όσον αφορά κάποιες εμπορικές συναλλαγές. Φυσικά αυτό είναι το, το στο μάλλον πιο σημαντικό υπό τη σημερινή συγκυρία ε, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα των επιχειρήσεων, γιατί καθυστερούν ε, οι πληρωμές και αυτές οι σημαντικές συνέπειες. Ε, είναι δυνατόν αυτό να οδηγεί σε πάυση πληρωμών και σε πτώχευση με τις κοινωνικές και άλλες συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό. Επίσης, η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι αυτή η οδηγία για την υπερημερία έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ. Γιατί αυτά είναι τα νομικά πρόσωπα τα οποία δημιουργούν την ε, μεγαλύτερη μεγαλύτερο κομμάτι της απασχόλησης στην κοινωνία. Έχει προχωρήσει η διαδρομή αυτού του σχεδίου οδηγία. Έχουμε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή σας, ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία Έχουμε κάποια σημεία προστριβής, διαφωνίες με εσείς, με, ως είναι αλήθεια. Και το Συμβούλιο έχει κάποιες ομάδες εργασίας που εξετάζουν αυτά τα σημεία. Νομίζω όμως θα καταλήξουμε σε ικανοποιητική λύση και ήδη έχουν αρχίσει επαφές άτυπες με τους ε, εισηγητές σας για να μπορέσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς να καταλήξουμε σε συμφωνία και να πάρει το δρόμο της η οδηγία. Επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι συναρμόδιες για το θέμα αυτό έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις τροπολογίας και ελπίζω ότι το πράγμα θα λάβει αίσιο τέλος. Τώρα, να σας πω κάτι άλλο το οποίο έχει σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ και πρώτα πρώτα έχουμε την πειρατεία παραποίηση προϊόντων εντός και εκτός της Ένωσης. Είναι κάτι το πάρα πολύ αρνητικό όσον αφορά τις επιχειρήσεις της καινοτόμες. Εκείνοι οι οποίοι πασχίζουν για περισσότερη καινοτομία. Αυτοί είναι που βοηθούν την απασχόληση, στην Ένωση και την οικονομική ανάπτυξη. Βεβαίως η παραποίηση είναι κίνδυνος και για την υγεία των πολιτών. Άρα θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για δημιουργικότητα, για καινοτομία και να κάνουμε κάτι όσον αφορά την παθολογία της, ε, ε, της, της αυτό το οποίο την, την, την πλήση, την πειρατεία. Οπότε, στο Συμβούλιο ήδη εγκρίναμε την ανακοίνωση της Κομισιόν επ' αυτού. Αυτό έγινε με ψήφισμα του Συμβουλίου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε επιτυχία την παραποίηση των προϊόντων και την πειρατεία. Επίση, εκφράζει την ικανοποίηση του Συμβούλιο, διότι το ισχύουν τα όσα είπαμε για παρατήρηση των εξελίξεων όσον αφορά τη πνευματική διοκτησία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική οδηγία. Επίσης, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για μια πολυμερή σύμβαση που θα βοηθήσει στην καταπολέμηση πειρατείας και παραπίεσης προϊόντων. Λέγεται άκτα αυτό το κείμενο και βέβαια λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες των εμπλεκομένων. Συνομιλούμε με κάποιες χώρες για να μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτή η συμφωνία. Λαμβάνουμε υπόψη τη θέση, τη δική σας, όσον αφορά το ψήφισμα για τις επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο της παραποίησης και έχουμε και κάποια πρόσφατα έγγραφα, όπως κάτι το οποίο βγήκε την περασμένη εβδομάδα πάνω σε αυτό. Πρόκειται για ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίνεται στην σύνοδό σας όπου και τονίζεται ότι είναι πάρα πολύ βασικό το να υπάρχει διαφάνεια στην καταπολέμηση πειρατείας και παραποίησης. Επίσης, εκεί, στο κείμενό σας, προβάλλεται τον ρόλο, τον σημαντικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκβαση αυτών των ε, διαπραγματεύσεων. Επίσης, εκτός από αυτά, πάλι για την πνευματική διοκτησία, θέλω να σας πω για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πολιτικά. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, γνωστό θέμα. Παρά το ότι έχει πολυετή διαδρομή, έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, αλλά όχι το κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Άρα, εάν μπορέσουμε να καταλήξουμε και μια συμφωνία, αυτό θα τονίσει πάρα πολύ την καινοτομία. Και γι' αυτό και το Συμβούλιο πρόκειται να εντείνει τους ρυθμούς εργασιών, ούτω ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Και γι' αυτό και αρχίσαμε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επιτροπό Μπαρνία να μπορέσουμε να δώσουμε μια όθηση στα πράγματα, να το διακυπηρεώσουμε το θέμα όσο γίνεται συντομότερα. Ακόμα περιμένουμε μια δικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οπότε και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα οποία ακόμη κρεμούν όσον αφορά το νομοθέτημα. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό θα έχει πλήρες συνομοθετικές αρμοδιότητες Και γι' αυτό και εμείς ως Προεδρία θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος μαζί σας. Εν κατακλείδη θέλω να πω κάτι για την νομοθετική πρωτοβουλία όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού. Και επ' αυτού ε, επ' αυτού έχουμε ένα σχέδιο οδηγίας που θα τροπήσει την οδηγία του 2008, την 116 λαμβάνω υπόψη τις προτάσεις σας, αλλά και συμφωνούμε με αυτό το οποίο προτείνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των ερμηνευτών, των εκτελεστών. Εάν θέλουμε να δώσουμε μια όθηση και κίνητρο στην καλλιτεχνική δημιουργία. Επομένως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε και αυτό το θέμα. Θα κλείσω τώρα, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η σημερινή συγκυρία. Είναι όμως και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι επίσης μια ευκαιρία για δημιουργικότητα. Αυτό το οποίο είπα προηγουμένως για τους δημιουργούς διότι υπάρχει οικονομική πίεση αλλά έχουμε τα μέσα αντιμετώπιση της οικονομικής πίεσης και το πρώτο μέσον και καλύτερο είναι η ιστορική αγορά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση, κάθε θεσμικό όργανο, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο όλοι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια συνένεση στο πώς η κρίση θα αποτελέσει ευκαιρία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει μπροστά της κάποιο εμπόδιο, το οποίο πάντοτε υπερπίδεσε και βγήκε πιο δυνατή από τη διαδικασία αυτή και είναι και αυτό το οποίο θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την ευρεία κάλυψη των θεμάτων. Ήταν σαφέστατα αυτά που είπατε. Υπάρχουν θέματα που αφορούν την ιστορική αγορά και βρίσκονται πραγματικά στην καρδιά της uh, αποστολή σας. Για μας ε, η εσωτερική αγορά είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά πιστεύω ότι πολλοί θησαυροί κρύβονται πίσω από αυτό που βλέπουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε, να κοιτάξουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπουμε και ελπίζω ότι και ο κύριος Μόντι και εμείς επεξεργαζόμαστε τα θέματα αυτά με μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να σας πω ότι στις 25 και 26 Μαΐου θα μας παρουσιάσει ο κύριος Μόντι κάποιες προτάσεις και ίσως θα ήταν καλό από κοινού με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συναντήσει τον καθηγητή, τον κύριο Μόντι, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο να σχολιάσουν, να κάνουν ερωτήσεις. Ο Κορέα Δεκάμπος, ο κύριος Φάμπ και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και άλλοι θέλουν να σας κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Κορέα Δεκάμπος είναι ο πρώτος και κατόπιν θα δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους και στον κύριο Άριας αν θέλει. Presidente, queria cumprimentar o Κύριε Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Τον ευχαριστούμε γιατί ο λαός αυτά μας ε, είπε αφορούν πάρα πολλές πρωτοβουλίες, ιδέες και προτάσεις οπότε επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε για το, κρυμμένο κόσμο, το κρυμμένο θησαυρό είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να το, να το προσέξουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ε, πολλές φορές όμως είναι σαν ε, δεν είναι αυτό το κρυμμένο κόσμο είναι παγόβουνο οπότε πρέπει να προσέχεις κανείς πάρα πολύ ε, αυτό το οποίο φαίνεται ότι γυαλίζουν θησαυρό, αλλά από κάτω είναι επικίνδυνο. Για να δούμε τώρα, για αυτό που είπατε όσον αφορά τι ε, υπηρεσίε και όσον αφορά την αξιολόγηση αυτή που είπατε ότι πρόκειται να, να γίνει. Ε, η αξιολόγηση δεν γίνει από το Συμβούλιο, θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για κάποιες δύσκολες, περίπλοκες οδηγίες και από πλευράς ιδεολογικής. Ε, αυτό ισχύει και για την οδηγία των ε, υπηρεσιών. Η εφαρμογή της είναι δύσκολη, χρειάζεται χρόνος. Για πέστε μας, πώς το βλέπετε. Μήπως πρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε την οδηγία, να, να, να βγάλουμε αυτό το στοιχείο το ιδεολογικό, το οποίο την έκανε αυτή την ε, οδηγία σε, σε κόκκινο πανί για πολλούς και μες στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου. Μήπως λοιπόν πιο εύκολα θα υλοποιήσουμε τα τη οδηγία των υπηρεσιών με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερη ερώτηση όσον αφορά με τα προϊόντα της φαρμακοβιομηχανίας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρμοδιότητα της Προεδρίας, αλλά η σχετική δέσμη, η νομοθετική, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος αλλά πρόκειται να συνεξετάσουμε και εμείς με την ε, Επιτροπή εκείνη ε, μια σχετική έκθεση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα παρπημένα φάρμακα της απομιμής φαρμάκων οπότε για πέστε μας θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται η ενημέρωση των ασθενών Είναι θέμα πάρα πολύ επίμαχο. Έχει, έχουν διφορούμενο, ε, έχουμε, μας έχει διχάσει ε, τις, τις με, μεγάλες πολιτικές ομάδες. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι δανειστές, κάποιοι πιστωτές, κάποιοι που έχουν κάποια ε, ε, οικονομική ισχύ. Πολλές φορές όμως αξίζουν και αυτή της προστασίας γιατί πολλές φορές και αυτοί όπως και ΜΜΕ υπό τη σημερινή συγκυρία έχουν πρόβλημα όσον αφορά τη, την πρόσβαση στις ε, αγορές χρήματος. Επίσης, ε, Θέλω, κάτι να σας πω για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και αυτό δεν είναι άμεση αρμοδιότητά σας. Πάντως, ε, είναι πάρα πολύ αξιόλογο το ότι έχετε την τόλμη να ασχοληθείτε με το δίπλωμα ευρεσιτεχνία που είναι κάτι που όλοι συμφωνούμε ότι εκκρεμεί ενώ θα πρέπει να εκπαιδευτεί εδώ και καιρό. Președinția spaniolă și-a început mandatul odată cu punerea în aplicare a tratatului. Η Προεδρία ξεκίνησε το πρόγραμμά της όσον αφορά την, το πρόγραμμα της Λισαβόνας. Έχουμε μια καινούρια επιτροπή και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η Ισπανική Προεδρία δεν έχει εύκολο έργο. Και εάν θέλουμε εδώ να παρουσιάζουμε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά αυτής της στρατηγικής. και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια στιγμή θα βγουν από την οικονομική κρίση και μόλις αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να ενδυναμώσουμε την εσωτερική αγορά. Πριν όμως γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία έχει μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα προς την ενσωμάτωση της κοινωτική νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια αφορούν άμεσα την οδηγία για, την, για τις υπηρεσίες καθώς και την αναγνώριση, την αναγνώριση. Και γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε για τις οδηγίες αυτές, για την οδηγία για τις υπηρεσίες παραδείγματος χάρη, να επεξεργαστούμε το θέμα με μια ειδική εργασία όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Το θέμα των ε, καθυστερημένων πληρωμών. Εδώ σαφώς και θα πρέπει να υπάρξει νέα προσπάθεια πειθαρχία για τις ε, αρχές των κρατών μελών. Αυτό θα έχει σαφώς πολύ θετικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας σε μια κοινή θέση όσον αφορά το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών. Και κάτι άλλο που συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μας, το θέμα της οδηγίας για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Εχθές συνεδριάσαμε σαν Επιτροπή και με την Επίτροπο την κυρία Ρέντινγκ μιλήσαμε για τις προσπάθειες που γίνονται όσον αφορά την προσπάθεια εξέβρεσης μιας κοινή θέσης για το θέμα αυτό της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σαφώς η οδηγία αυτή δεν θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και θα χρειαστεί άλλο ένα εξάμεινο πριν βρεθεί κάποια λύση ικανοποιητική για όλους αλλά θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικό για την Ισπανική Προεδρία να στηρίξει τεχνικές συζητήσεις ε, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ όσον αφορά την πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρυστεχνίας, γιατί το θέμα αυτό το συζητούμε πολύ καιρό και τίποτα δεν έχει γίνει. Ο κύριος Άριας Βερνιού, Τριανταφυλλίδης και Έγκστρομ. Ο Υπουργό θα φύγει στι 4. Σα παρακαλώ πολύ λοιπόν να είστε σύντομοι και ακριβεί στι ερωτήσει που κάνετε. Uh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και θα ήθελα να σας πω ότι κάτι δεν το αναφέρατε. Την οδηγία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Πρόκειται για κάποια οδηγία που την έχουμε στήσει πολλές φορές και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το άριστο ή το χείριστο γιατί θα πρέπει να δούμε άπαξ και ενταχθεί στην εσωτερική νομή τάξη να ισχύει για όλες τις χώρες της Ένωσης. Και έτσι, από την άλλη μεριά, αλλού θα ανέβει ο πύχης, αλλού θα κατέβει αναλόγω το τι ισχύει για τους καταναλωτές στην κάθε χώρα. Άρα, σας ρωτώ, πώς βλέπετε αυτό το προβληματάκι όσον αφορά τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο. Εκτός αν θεωρήσουμε ότι θα βάλει πολύ ψηλά τον πύχη η οδηγία αυτή, τι θα γίνει στην Ισπανία. Θα γίνει η ένταξη στο εργοδίκιο. Συμφωνώ και συζητήσαμε προηγουμένως με τον ε, Υπουργό ότι θα μας μιλήσει ενδεχομένως και για τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά θα επικεντρωθούμε κυρίως στην εσωτερική αγορά. Η κυρία Βενίου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό και την Προεδρία γιατί είστε πολύ παρόντες στις επιτροπές μας και όχι μόνο στο Στρασβούργο. Ήδη έχουμε συνεργαστεί και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεχίσουμε. Τι χαρητήρια λοιπόν. Μιλήσαμε και εμείς με τον Μάριο Μόντι όσον αφορά τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς και είδαμε από το 2005 πως οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή προσπάθεια δεν τους προστατεύει πλέον και ότι απομακρύνεται από τους αρχικούς στόχους. Το θέμα της οδηγίας για την υπηρεσία, για τις υπηρεσίες πρέπει να μας οδηγήσει σε μια ανάλυση και πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες για να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες βάσει των υπηρεσιών κοινής ωφελίας. Εγώ εργάζομαι σήμερα για μία οδηγία η οποία έχει κατά κάποιο τρόπο σταματήσει. Πρόκειται για την υπηρεσία, για τις ε, υπηρεσίες υγείας σε διεθνωριακό επίπεδο. Υπάρχει επίσης και όλος ο τομέας της ε, λεγόμενης οικονομίας αλληλεγγύης. Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν στους τομείς αυτούς και η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών μπορεί να βελτιωθεί. Το ερώτημα λοιπόν που σας κάνω είναι, επειδή θα ακολουθήσει η Βελγική Προεδρία, πιστεύετε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, έτσι ώστε και να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά, αλλά και να δουν με καλύτερο μάτι οι Ευρωπαίοι πολίτες την εσωτερική αγορά. Κάτι που σήμερα δεν το αναγνωρίζουν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό για τις πληροφορίες που μας έδωσε για όλα αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν τους επόμενους μήνες. Μας μίλησε για τις προσπάθειες του καθηγητή του κ. Μόντι για να επαναφέρει στο προσκήνιο την ιστορική αγορά. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση και εμείς ε, πρέπει να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Ο Υπουργός στην παρουσίασή του μίλησε για την δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής υπηκότητας. Τι ακριβώς εννοεί. Οι πολίτες θα γίνουν Ευρωπαίοι καταναλωτές είτε θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης γιατί ωραίο είναι να έχουμε μια εσωτερική αγορά η οποία εργάζεται με μεγάλη ακρίβεια σαν ελβετικό ρολόι αλλά το θέμα είναι βελτιώνοντας τα πράγματα να επωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν θέλω να ακούσω λοιπόν την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τριανταφυλλίδη. Τέλος ο κύριος Έγκστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για το ψήφισμα που πέρασε από την Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλήσατε για τη διαφάνεια και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι προτίθεται να κάνει συγκεκριμένα η Ισπανική Προεδρία έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει τα στοιχεία και τα έγγραφα εγκαίρως όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο του συναδέλφου, για όλε αυτέ τις ερωτήσει. Και θα δώσω το λόγο στον Υπουργό, έτσι ώστε να σχολιάσει και να απαντήσει. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ο Πρόεδρος. Ο Γιώργος Υπουργός, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αρχίσω τις ε, απαντήσεις συμφωνώντας με αυτό το οποίο είπε τόσο ξεκάθαρα ο πρώτος Επιτροπής ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία Συμβουλίου και τη Κοινοβουλευτική επιτροπή, σας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα βήματα προ τα εμπρό. Γι' αυτό θέλω να πετύχουμε, δηλαδή την ε, τόνωση, την όθηση στην εσωτερική αγορά. Αυτό το κόσμο, το θησαυρό τη Ένωσης. και θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο, πιο, πιο ορατός, πιο προβελμένος αυτός ο θησαυρό. Οπότε, εάν υπάρχουν κάποιες πλευρές αυτής της ε, ιστορικής αγοράς, κάτι το οποίο έχει, έχει θολώσει, θα πρέπει να δώσουμε την, την έγκλη που είχε, να λάμπει και πάλι αυτός ο θησαυρό, αυτό το κόσμημα, από τις ακτίνες του ήλιου, του ήλιου των Βρυξελών. Όποτε έρχομαι, πετυχαίνω ήλιο εδώ. Οπότε θα πρέπει αυτό ο θησαυρό τη εσωτερική αγορά να είναι δυνατόν να αναδειχθεί αυτό και όλε του οι δυνατότητε και να προβληθεί προ του Ευρωπαίου πολίτε. Ακριβώ όπω είπε και ο κύριο Τριανταφυλλίδη. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις που έγιναν σε σχέση με την έκθεση Μόντι και το ότι πρόκειται έτσι να δούμε ποιες είναι οι νέες προοπτικές στην ιστορική αγορά για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε αυτή την πρόταση για ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο στο μέλλον. Και αυτό θα έχει κομβική σημασία στην εσωτερική αγορά. Επίσης, πολύ έλαβαν το λόγο και θα πρέπει να σας πω εκ μέρους του Συμβουλίου ότι η Κομισιόν, ο πρόεδρος Μπαρός ζήτησε να συνταχθεί αυτή η έκθεση όμως και εμάς μας ενδιαφέρει θα τη μελετήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα αξίζει πάρα πολύ γιατί γνωρίζουμε ποια είναι η διαδρομή του Μάριο και ξέρουμε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά σε τέτοια πράγματα και ε, ήδη αυτό που σαν προκαταβολή μας, μας εξήγησε την περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ αξιόλογο οπότε γι' αυτό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πάρα πολύ δημιουργική συζήτηση στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού και Ανταγωνιστικότητας. Επίσης, πρόεδρε, θεωρήστε ότι σας προσκαλώ στη συζήτηση εκείνη που θα γίνει στο Συμβούλιο. Και θέλουμε για τη δική σας άποψη, τη χρειαζόμαστε, γιατί είναι στατική σημασία στο ζήτημα αυτό. Αλλά είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά η ιστορική αγορά, είναι θέμα στατική σημασία για την Ένωση για την Ένωση του 21ου Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε από κοινού τα τρία θεσμικά όργανα. Οπότε και πάλι σας λέω Πρόεδρε, σας προσκαλώ, ελάτε να συζητήσουμε με τον Μάριο Μόντι. Περιμένουμε πώς και πώς να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Επίσης, κάποιοι έλαβαν τον λόγο και μίλησαν για την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Ο, ο κύριος Κάμπος και άλλοι μίλησαν για την οδηγία αυτή η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η ύψιστη της σημασίας τη θεωρώ και είναι τόσο σημαντική τόσο πολύ βρίσκεται στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής, της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς που μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνω και πέρα από ιδεολογικές θεωρήσεις που θα περιόριζαν το βεληνικές της. Γι' αυτό σας λέω κύριε Κάμπος ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε όσο γίνεται περισσότερο το να μπορέσει αυτή η οδηγία να διαπνέει κάθε δραστηριότητα και όσο γίνεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να αποκτήσει η δραστηριότητα αυτή η οικονομική μία ισχύ πάρα πολύ σημαντική και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Γιατί μιλούμε για απορρίθμιση στον κλάδο των υπηρεσιών. Μιλάμε για περισσότερες δυνατότητες μιλούμε για άρση κάποιων ολιγοπολίων που υπάρχουν σε διάφορα Δηλαδή πρόκειται για ένα μετασχηματισμό που φέρνει αυτή η οδηγία και για αυτό και πολλοί αντιστέκονται στην εφαρμογή της. Όπως ξέρουμε αλλού έχει, αλλού δεν έχει ε, εφαρμοστεί και αυτό γιατί κάθε φορά που κάποιος προτείνει κάτι αισιόδοξο πάντοτε βρίσκει κάποιους να θέλουν να του βάλουν τροχοπέδι και άλλωστε πάντα έτσι ήταν. Ε, κάνει βήματα προς τα μπρος η Ένωση, απ' την άλλη υπάρχουν τάσεις ε, πανεθνικοποίησης και γίνεται μετά η υπέρβαση αυτών των αντιστάσεων για αυτών των ε, δύο. Άρα και εμπροκειμένα θα υπάρξουν κάποια τέτοια εμπόδια. Ήδη φάνηκε αυτό πριν, όπως είπε ο κ. Βουλευτής Κορέγια, να φάνηκε το, το, πώς θα υπάρχουν οι αντιστάσεις. Όμως ή είμαστε αποφασισμένοι η Ένωση και η Ισπανική Προεδρία. Όπως και εσείς ε, είπατε, θέλουμε να γίνει η μεταφορά αυτής της οδηγίας στο δίκαιο και επομένως να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει για να υπάρχει η αναγκαία μεταρρύθμιση και να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να φτάσουμε σε πιο υγιή και σταθερή και ποιοτική οικονομική ανάπτυξη. Γιατί όλοι στο 2020 έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά και βασικός άξονας είναι η οδηγία αυτή. Τώρα, κάποιοι άλλοι ανέφεραν στην οδηγία για την καθυστέρηση των πληρωμών. Είναι προτεραιότητα για μας αυτή η οδηγία για την υπερημέρεια. Έτσι με αυτή την οδηγία θεωρούμε ότι θα ευνοήσουμε, θα, θα δημιουργήσουμε θετικό κλίμα για τις ΜΜΕ. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σαφές, πριν είναι κάτι το οποίο όλες τις ΜΜΕ θα τις καλύψει, αλλά ιδίω από όλες τις επιχειρήσεις που θα καλύψει, κυρίως τις, τις ΜΜΕ, γιατί αυτές έχουν μικρότερες ε, αντιστάσεις στη δύσκολη συγκυρία. Οπότε γι' αυτό και θεωρούμε ότι πρόκειται για οδηγία η οποία είναι πάρα πολύ απαραίτητη και θα πρέπει και αυτή να εφαρμοστεί όσο γίνεται συντομότερα. Και γι' αυτό το λόγο επίσης όπως είπε ε, ο κύριος Μπέστη θα πρέπει η οδηγία αυτή να σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό επιδιώκουμε. Φυσικά υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία διαφωνίας όπως ε, ε, όσον αφορά τη ρύθμιση της διαφοράς μεταχείρισης μεταξύ δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων ή κάποιες ε, κυρώσεις για, για την αδυναμία πληρωμής. Θα πρέπει νομίζω όμως αυτές οι διαφορές μας να γεφυρωθούν να μπορέσουμε να φτάσουμε επομένω με αίσιο τρόπο στην ε, ψήφιση που θα γίνει στις 8 Απριλίου στην Επιτροπή σας και αυτό το θέλει πάρα πολύ η Ισπανική Προεδρία γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό κείμενο οπότε και θα πρέπει αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες να θεωρήσουμε ότι φέρουν πιο κοντά στην Ένωση τους ε, πολίτες ε, γιατί έτσι φαίνεται, προβάλλεται η πρακτική χρησιμότητα της Ένωσης. Και γι' αυτό και θα πρέπει πάνω σε αυτά να, να, να επιμένουμε περισσότερο, θα πρέπει να είμαστε πιο διεκπαιδευτικοί ακριβώς. Παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων είναι η οδηγία τη υπερημερία. Επίση, κάποιοι άλλοι αναφέρθηκαν επανειλημμένα στο θέμα τη ευρεσιτεχνία τη κοινοτική. Σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια που εμεί τάξαμε σαν προτεραιότητα την ε, κοινοτική ευρεσιτεχνία. Έτσι, θεωρούμε ότι μπορούμε τελικά να φτάσουμε σε κάποια συνένεση όσον αφορά την ευρεσιτεχνή αυτή, θέμα το οποίο έχει μπλοκαριστεί τόσο χρόνια. Άρα θα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην υλοποίηση της ιδέας αυτής γιατί έτσι θα μας προσδώσει πάρα πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα σε κάθε συνάντηση με επιχειρηματίε, με οικονομικού παράγοντε, πάντα, πάντα, πάντα βγαίνει αυτό το θέμα, ε, πάγιο αίτημα. Γιατί θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία που υπάρχει σήμερα, ε, η ευρεσιτεχνία του Μόναχου, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, αναποτελεσματικό και άρα επομένω θα πρέπει να θυμηθεί πρόοδο. Και ακριβώ γι' αυτό και επεξεργαζόμαστε το θέμα, συνεργαζόμαστε συχνά, στενά με τον αρμόδιο επίτροπο που είναι ο κ. Μπαρνιά. Για τους καταναλωτές τώρα. Προστασία καταναλωτή. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκατε. Μπέσντι, Άριας. Κοιτάξτε, Δεν είπα τίποτα γιατί θεώρησα ότι ήδη το έχετε συζητήσει. Ευχαρίστως όμως να σας πω σχετικά, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και έμεσα να θίξω και κάτι άλλο που αναφέρθηκε. Ποιος ήτανε? Ο κύριος Τενταφυλίδης. Διότι αναφέρθηκε στο πόσο κοντά, στο πόσο ενταγμένη θεωρούμε ότι είναι ε, η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι στην εσωτερική αγορά. Πόσο κοντά είναι, γιατί βεβαίως και είναι πολύ σημαντική διάσταση της ζωής του καθενός στην Ευρώπη η κατανάλωση επομένω. Εάν έχουμε εδώ κάποιες ανισορροπίες, εάν έχουμε κατάχρηστες στους θέσει. Βεβαίω και αυτό παραβλάπτει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του Ευρωπαίου, του καταναλωτή. Προβλέπει σχετικά η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Έχουμε επίσης τον χάρτη, τη χάρτα των δικαιωμάτων των θεμελιωδών που ρυθμίζουν τα σχετικά. Και αυτό βέβαια με τίποτα δεν ε, παραβλάπτει, δεν συρρυκνώνει τη σημασία τη ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αναπόσπαστο τμήμα των, των, δικαιωμάτων του, ε, του Ευρωπαίου, το δικαίωμα του καταναλωτή και είναι κάτι το οποίο φυσικά παραπέμπει στο πότε και αν υπάρχει ανισορροπία και ανισότητα μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή. Οπότε ε, θα πρέπει κανείς, αν την αρμοδιότητά του, να επαναφέρει την ισορροπία, την δέουσα μεταξύ παραγωγού, αγοράς και καταναλωτή. Γι' αυτό και εμεί θέλουμε να προχωρήσει η οδηγία αυτή που προβλέπει για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Οπότε θα γίνει πιο εύρυθμη και η οδηγία τη εσωτερική αγορά Έχει να κάνει και με το δικαίωμα στην ενημέρωση και πληροφορία. Επίσης την επιστροφή των χρημάτων όταν έχουμε περιμερή, περιμερή εκτέλεση συμβάσεως τι θεωρείται καταχρηστική ρήτρα, όλα αυτά προβλέπονται εκεί γιατί είναι δικαίωμα του καταναλωτή αντίστοιχα. Οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς θα βρούμε μια ισόρροπη λύση μεταξύ των δύο αντιρρόπων συμφερόντων που θέλουμε να ρυθμίσουμε στην ε, οδηγία αυτή. Δηλαδή, πλήρη εναρμόνιση των ε, σχετικών νομοθεσιών της Ευρώπης και από την άλλη μεριά η άλλη τάση που λέει το να ελαχιστοποιηθεί, να γίνει, να υπάρχει μικρότερη δυνατή ε, εναρμόνιση. Εμείς θέλουμε να συμφωνήσουμε σε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο αντιρρόπων τάσεων. Και γι' αυτό και πρόκειται να το εντάξουμε αυτό το θέμα ως σημείο συζήτησης 25 26 Μαΐου. Και έτσι να αποκτήσουμε μια πρώτη ιδέα που θα κατευθυνθούμε με ένας να γίνει. Για να πάμε προς μια συνένεση και συμφωνία και να δούμε πώς θα μπορέσουμε πιο συχνά να τα λέμε εδώ με τη δική σας επιτροπή και έτσι να διευκολυνθεί η σύναψη κάποια συμφωνία. Όχι, δεν είναι αυτό που είπατε κύριε Άρια. δεν θα γίνει αυτό όντω στην Προεδρία μας, δεν θα ολοκληρωθεί, αλλά Πάντω. θέλουμε αυτή η οδηγία να ολοκληρωθεί κατά κάποια στιγμή ε, όσο έχουν την Προεδρία οι χώρες τη Τρόικας που είπαμε. Βέλγιο, Ουγγαρία, Ισπανία. Κάποια άλλα συγκεκριμένα θεματάκια όπως το ζήτημα των ε, φαρμάκων για το που μίλησε ο κύριο Κορέγια. Είναι προτεραιότητα αλλά όχι τόσο. Και δεν είναι ότι, δεν ότι εμεί δεν θέλουμε αυτό το θέμα κατά προτεραιότητα να διεκπαιρεωθεί, είναι ότι υπάρχουν, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν διαφωνίε. Ένα σωρό κρατημέλη, 20 κρατημέλη. Δεν θεωρούν ότι αυτό είναι θέμα προτεραιότητα σήμερα. Οπότε, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να κάτσει και να ξαναζυγίσει αυτή την πρόταση, ούτω ώστε να έχουμε κάποιο χαρτί πορεία για το θέμα αυτό. Τώρα όσον αφορά την φαρμακοεπιτήρηση, αυτό πάει καλά. Θεωρούμε ότι θα υλοποιηθεί σε πρώτη ανάγνωση αυτό που θέλουμε. Έχουμε βέβαια κάποια τεχνικά θεματάκια με την ε, επιτροπολογία, αλλά τα έχουμε βρει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό. Συμφωνεί επομένως ε, και η Ισπανική Προεδρία ότι έτσι μαζί θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Νομίζω ότι κάλυψα σχεδόν όλες Τι ερωτήσει. Α, η κυρία Βεργό. Σε για κάποιε διασυνοριακές υπηρεσίες και συμφωνώ μαζί τη. Εδώ φυσικά και υπάρχουν δυνατότητες απασχολησιμότητας, υπάρχουν δυνατότητες πάρα πολύ μεγάλες που υπάρχουν, αλλά θα πρέπει αυτό να είναι μια προτεραιότητα που να τάξουμε εμείς και οι επόμενε δύο προεδρίες, Ούγγρη και Βέλγια. Πάνω σε αυτό που είπατε. Γιατί ε, ακριβώ είναι πάρα πολύ σημαντική η αγορά των ε, υπηρεσιών. Και γι' αυτό και θα πρέπει και η σχετική οδηγία να εφαρμοστεί, να, να σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε, μοιραία ναι, και αυτό δεν είναι δική μας ε, προτεραιότητα και στόχος. Νομίζω απάντησα στις ε, ερωτήσεις σας και επαναλαμβάνω Πρόεδρε. Σας προσκαλώ να έρθετε να συζητήσουμε για την εσωτερική αγορά. Και έτσι να αρχίσει μια διαδρομή συνεργασίας μεταξύ μας. Ακριβώς για τα αυτά τα στρατηγικά θέματα που σε αυτή τη φάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να διεκπαιρεωθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της ε, διαφάνειας ενδεχομένως δεν απαντήσατε. Ναι, ναι, θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια όσον αφορά, συμπληρωματικά όσον αφορά την προσβασιμότητα των εγγράφων. Ε, είμαστε σε επαφή και με την Επιτροπή βεβαίω ακριβώς για να τροποποιηθεί ο κανονισμός όσον αφορά την προσβασιμότητα των εγγράφων. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι βεβαίω είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε ε, στην διοργανική διαθεσμική ε, ομάδα εργασίας που νομίζω ότι θα συνεδριάσει τον μήνα Μάιο έτσι ώστε να ακολουθήσουμε και την γραμμή που προτείνει το Κοινοβούλιο. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Υπουργέ γιατί ε, πραγματικά απαντήσατε με διεξοδικό τρόπο σε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε επίσης ε, και για την ε, πρόσκληση να συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο στη συζήτηση με τον ε, καθηγητή κύριο Μόντι. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψουμε όλοι μαζί και βεβαίως με τον σαφή ενθουσιασμό που δείξατε για την ενιαία χώρα τα πράγματα είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουν καλύτερα και πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ που δείχνετε τέτοιο, τόσο μεγάλη ενεργητικότητα ε, και είμαστε βέβαιοι ότι ε, μέσω ημών το Συμβούλιο θα κινηθεί γρήγορα έτσι ώστε η οδηγία στην οποία αναφερθήκαμε να ενσωματωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα για το μέλλον, για την Προεδρία σας ε, Ξέρω ότι σε πολλά θέματα τα οποία είναι αρκετά προβληματικά όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών έχετε μεγάλο ενθουσιασμό και δουλεύετε από πολύ κοντά. Ε, γνωρίζουμε ότι θα είστε και στο Στρασβούργο λίγο πριν ολοκληρωθεί το εξάμεινο της Προεδρίας σας. Οπωσδήποτε σας περιμένουμε, οποτεδήποτε ε, ε, θελήσετε και πρέπει να σας πω ότι η δουλειά σας έχει πολύ θετικό πρόσημο για μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Uh, um, uh, Πρόεδρος, νομίζω ότι τώρα μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε με τις εργασίες του απογεύματος. Έχουμε μερικά σημαντικά θέματα, σημαντικές γνωμοδοτήσεις να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ολοκλήρωση εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο συνάδελφος ε, Παύλο Αρίας Ετσεβερία θα κάνει την παρουσίαση και έχουμε και τον κύριο Κάμπος, ε, σκιώδη συγητή. Ε, είστε και εσείς ε, κυρία Ένστον. Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν και άλλον σκιώδη συγητή. Μερικοί λείπουν και ο κύριος Σαβίνη λείπει. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Αρίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι εισηγητής σε αυτό το έγγραφο ίδιας πρωτοβουλίας σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και μέσα στα πλαίσια της ε, ολοκλήρωσης αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα. Γνωρίζουμε αυτήν την επανάσταση ε, χωρίς προηγούμενο που έφερε το διαδίκτυο. Άλλαξε συλλήβδην το παγκόσμιο εμπόριο το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει, την, ε, δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, δίνει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στους ε, ε, τους καταναλωτές της Ευρώπης και επομένως έχει ως αντίκτυπο τον, την μεγάλη ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Απ' την άλλη πλευρά έχουν αυξηθεί και οι δυνατότητες και προσφοράς και επιλογής από πλευράς των καταναλωτών οι επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, ε, δρούν μέσα στα πλαίσια αυτού του εμπορίου μπορούν να φτάσουν μέχρι πελάτες και καταναλωτές τους οποίους με, καμία, με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσαν, στους οποίους δεν θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση με διαφορετικές συνθήκες. Πρόκειται για ε, μια αγορά η οποία διαρκώς διευρύνεται. Αγοράζουμε τα ηλεκτρονικά εισιτήριά μας ε, για το, το αεροπορικά μας ταξίδια, ε, πληρώνουμε ή κλείνουμε τα ταξίδια μας, τα ξενοδοχεία μας, τα εισιτήριά μας για θεάματα, θέατρα κλπ. Πάντως ε, υπάρχει και μία σειρά προσκομμάτων που θα πρέπει να αρθούν έτσι ώστε πραγματικά να αρθούμε στο ύψος ε, της νέας οικονομικής πραγματικότητας και της νέας ε, παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με το θέμα αυτό και στις 21 Ιουνίου του 2007 βασιζόμενο στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της κυρίας Ροϊτόβα ασχολήθηκε με το θέμα της εμπιστοσύνης των πολιτών ε, όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική αγορά. Ε, τον Οκτώβριο επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, έκανε ανακοίνωση ε, του κανονισμού σχετικά με το διασυνοριακό εμπόριο online και προτάθηκαν μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχει επίσης ε, το, η πρόσφατα δημοσιευθήσα τον Οκτώβριο του 9 μελέτη σχετικά με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και το αντίκτυπο ε, στον εμπορικό κόσμο αλλά και στους καταναλωτές. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει αυξηθεί ε, αναλογικά αντίστοιχα η χρήση του διαδικτύου όσον αφορά το, τις συναλλαγές ε, online διότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών ε, και φόβος ότι η ποιότητα δεν θα είναι αυτή που, που επιθυμούν κτλ. Ε, αυτή τη στιγμή επίσης προσκόμματα στην ολοκλήρωση της ε, ηλεκτρονικής αγοράς, της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν ε, κατακαιρματισμός των, ο κατακαιρματισμός των αγορών, η επιβολή φόρων που είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η ελευθερία συναλλαγών, η ελευθερία ανταλλαγών υπηρεσιών και αγαθών αποτελεί ε, μία από τις βασικές ελευθερίες και επομένως έναν από τους πυλώνες πάνω στον οποίο στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένα οπλοστάσιο ομοιογενών ε, κανόνων που θα διέπουν την εμπορική δραστηριότητα μέσω του διαδικασίου έτσι ώστε να επιτρέπει στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα αυτό να είναι ανταγωνιστικές χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία ε, θα αφορά όμως και ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη ε, και των επιχειρήσεων αλλά και των ε, καταναλωτών, ε, να αυξήσουμε λέω την εμπιστοσύνη τους ε, στο εμπόριο online. Να δημιουργήσουμε λοιπόν μία ενιαία οδηγία για ολόκληρη την Ευρώπη. Να υπογραφούν διεθνείς συμφωνίες οι οποίες θα διασφαλίσουν το ότι οι επιχειρήσεις δεν θα χάνουν ανταγωνιστικότητα όταν θα βγαίνουν εκτός των συνόρων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό έτσι ώστε να μην το καλύπτει ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ε, πρέπει να πούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει το στοιχείο αυτό βασικό στοιχείο και της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ο πρόεδρος ε, της ε, Κομισιόν, ο Χουάν Μανουέλ Μπαρόσο, αναφέρθηκε ε, στο θέμα αυτό σαν ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Επομένως, θα πρέπει να δουλέψουμε και αυτό σε, πολλές, σε πολλαπλή βάση. Πρώτον, είναι απαραίτητο να έχουν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης ποιοτική πρόσβαση στο ε, διαδίκτυο έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε συναλλαγές ε, δια του διαδικτύου. Επομένως, στις χώρες αυτές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν είναι ικανοποιητικές, αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουν την ποιότητά τους και αυτό θα αποτελέσει ήδη ένα μεγάλο βήμα προς τα ευρώς. Δεύτερον, θα πρέπει να ξεπεραστεί ο Τη ε, της αγοράς ε, online έτσι ώστε να ε, προχωρήσει πραγματικά το διασυνοριακό εμπόριο διότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε υπηρεσίες οι οποίες δεν προτείνονται ή δεν είναι διαθέσιμες για το ε, διασυνοριακό ε, εμπόριο ή ε, ότι σε κάποιες συναλλαγές δεν γίνονται δεκτοί αγοραστές από ορισμένες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί σίγουρα το άρθρο 20β της ε, οδηγίας ε, για τις υπηρεσίες που απαγορεύει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση και οποιαδήποτε διαφοροποίηση των αγοραστών πελατών. Τρίτον, θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Αυτό ε, θα, αυτό θα πρέπει να αφορά όχι μονάχα την ώρα ή τη στιγμή της υπογραφής της ε, σύμβασης, αλλά θα πρέπει με τον ίδιο κανονισμό να διευθετηθούν και να αποσαφινιστούν και ζητήματα τα οποία αφορούν τη σχέση αγοραστού ε, πελάτου και είναι ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί και ο συνάδελφος κ. Σουάμπ. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ε, αγοραστών στις συναλλαγές online. Δεν εμπιστεύονται αυτή την αγορά πάρα πολλοί οι αγοραστές, πάρα πολλοί καταναλωτές για πολλούς λόγους. Γιατί φοβούνται ότι θα τους στήσουν παγίδα, γιατί φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν το αντικείμενο της αγοράς τους εάν δεν τους ικανοποιεί. Επομένως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας, ε, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα σωστής εποπτείας του διαδικτύου, αλλά φυσικά να υπάρξουν και οι απαραίτητες για την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών εκστρατείες πληροφόρησης για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα Πέμπτο, θα πρέπει να ε, υπάρξουν πρωτοβουλίες για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν ε, να ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες φοβούνται να ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη τα νομοθετικά φορολογικά συστήματα ε, μπορεί να διαφέρουν και να τους δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Επομένως όλο αυτό το πλαίσιο είναι ε, δύσβατο, είναι ακριβό και πολλές φορές ακατάληπτο. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, ανοίξουν οι δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις να ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω ας πούμε απλούστευσης των διαδικασιών σχετικών με το ΦΠΑ ε, η επίλυση πρακτικών προβλημάτων σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτασίας ε, η ε, με πάυση του συστήματος όπου καμιά φορά χρειάζεται μια επιχείρηση να πληρώσει πολλές φορές για το ίδιο πράγμα σε διαφορετικές χώρες κτλ. Έκτο, θα πρέπει να αυξηθεί η ασφάλεια της χρήσης ε, του διαδικτύου. Θα πρέπει να υπάρξουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μηχανισμοί ε, που θα προστατεύουν τους ανήλικους ε, κατά την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και αυτό θα πρέπει να αφορά και την, ε, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ε, ε, και τα chat rooms κτλ. Ε, πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να βελτιωθεί και όλη η κατάσταση σχετικά με, το, με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, αναπτύξουμε και να συζητήσουμε περιττέρω σχετικά με τις ε, ιδέες αυτές ε, που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο και βεβαίως είμαι στη διάθεση όλων να συζητήσουμε και να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε εδώ τον, ε, κύριο, τον κύριο καθηγητή Κορέας Δεκάμπος, έχουμε τον κύριο Κρότσμαν. Νομίζω ότι εγώ θα μιλήσω εξ με της ομάδος μου, γιατί δεν είναι παρόν ο, ο αντίστοιχος ε, σκιώδης. Και πρέπει να σας πω ότι είναι και πυκνές οι γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα. Ήρθε πραγματικά με μεγάλη δύναμη η Κομισιόν σήμερα. Έχουμε και παλιούς γνώριμους από την συζήτηση που ξεκινήσαμε για την οδηγία ε, για τις ε, υπηρεσίες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, της Επιτροπής. Ο καθηγητής Κορία Ντεκάμπος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν εξαιρετική η συμβολή του στην πρόθεση της, ε, του θέματος αυτού. Πιστεύω ότι ανοίγεται μπροστά μας μια εξαιρετική ευκαιρία. Ένα νέο πεδίο λοιπόν ανοίγεται μπροστά μας. Μέχρι τώρα φτάσαμε, μέχρι εδώ που φτάσαμε, χωρίς ε, ιδιαίτερη νομοθεσία. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον θα πρέπει να ενεργήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, θα ήθελα να κάνω μερικά θετικά και μερικά αρνητικά σχόλια. Είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε ε, πληροφόρηση ε, γνωρίζομαι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι συναλλαγές ε, μέσω διαδικτύου. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι και πιο σημαντικό να ε, προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο τον καταναλωτή. Επίσης για μικρές αγορές, ε, ας πούμε είτε προϊόντα ε, τεχνολογίας πληροφορίας, είτε αγορά βιβλίων, μικρών ενδυμάτων, ε, ή εισιτηρίων θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια αρνητικά. Οι γεωγραφικές ασυμμετρίες όσον αφορά την διεύρυνση ε, και την διάχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανισορροπία ε, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη επίσης οι χρήστες ε, του διαδικτύου ξεπερνούν το 80% ε, και αυτοί οι άνθρωποι ε, πραγματικά είναι δυνάμοι αγοραστές χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά σε μερικές περιπτώσεις δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους αγορές γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί. Π.χ. Ε, ο μη εναρμονισμένος φόρος προστιθέμενης αξίας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα για να ε, μπορέσει να ε, λειτουργήσει το σύστημα πρέπει κανείς να ανοίξει λογαριασμό στην χώρα παράδοσης, τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης το cash on delivery και αυτό μας προκαλεί πολλά προβλήματα. Ε, πρόκειται για τις αγορές με αντικαταβολή που έχουν οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό παραπώνων. Ε, πάντως, όπως είπε και ο εισηγητής, το θέμα είναι ε, όχι ιδιαίτερα περίπλοκο, είναι εύκολο να καταλάβουμε τις δυνατότητες που μας ανοίγονται για το μέλλον εάν ανοίξουμε αυτή την πόρτα που μέχρι τώρα είναι κλειστή. Ο κύριος Κρόιτσμαν, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχει μας έχει πει ο εισηγητής, μόλις τον ακούσαμε, πού είναι τα προβλήματα. Εγώ λέω ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης και για αυτούς που προμηθεύουν το εμπόρευμα και, αυτούς που, σε αυτούς που αγοράζουν το εμπόρευμα. Για την αγορά ε, ας πούμε εισιτηρίων Ε, ξέρουμε ότι δίνουμε τον αριθμό της κάρτας μας. Επομένως, ε, ε, αυτό δείχνει ότι έχουμε εμπιστοσύνη σε ορισμένες μορφές, ακόμα και όταν πρόκειται για αγορά διπυρωτικών εισιτηρίων. Ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα πράγματα λειτουργούν πάρα πολύ καλά και ότι μέσα από γρήγορο ταχυδρομείο μας στέλνονται ε, αμέσως τα αντικείμενα τα οποία έχουμε αγοράσει κτλ. Τώρα ε, τι γίνεται, μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα. Ε, φτάνει το προϊόν και έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή έχει ήδη πληρωθεί έχει πληρωθεί μέσω της πιστοτικής κάρτας ένα αντικείμενο ε, το οποίο τελικά ε, είναι προβληματικό και εκεί αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι σαν καταναλωτές ότι είμαστε προστατευμένοι μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει ε, το ε, αντικείμενο το οποίο έχει, έχουμε αγοράσει και θα είναι σε καλή κατάσταση. Ε, επίσης ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστραφεί ε, τότε θα πρέπει επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες έτσι όπως ε, ορθά προβλέπονται από τον νόμο κτλ. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πελατών. Γιατί διαφορετικά, εάν δεν έχουμε δηλαδή εμπιστοσύνη, τότε μειώνεται όλο και περισσότερο, συρρυκνούται όλο και περισσότερο η αγορά. Με την έννοια ότι ε, πιθανοί αγοραστές οι οποίοι ε, θα μπορούσαν να προσθεθούν εις ε, τους αγοραστές μιας επιχείρησης, προϊόντων μιας επιχείρησης δεν τολμούν να αγοράσουν ε, τα προϊόντα αυτά γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, όσον αφορά επίσης την δυνατότητα παραβίαση προσωπικών δεδομένων, όσον αφορά τα στοιχεία πληρωμής κτλ. Αυτά νομίζω ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο αύριο. Λείπει λοιπόν η απαραίτητη εμπιστοσύνη για όλα τα άλλα θέματα. Θα βρεθούν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν. Όπως παραδείγματο χάρη η εξασφάλιση των πληρωμών με ηλεκτρονικό τρόπο κτλ. Το βασικότερο και αυτό από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, το καθοριστικό, είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης, κλίματος εμπιστοσύνης, καθότι όταν κάποιος παραγγέλνει ένα προϊόν, Ξέρετε ότι μέχρι να το παραλάβει και να σιγουρευτεί ότι είναι σωστό υπάρχει μεγάλη, μεγάλη αβεβαιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Έγκστρομ, σαφώς και το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη. Είναι ένα από τα έργα που σαν πολιτικοί θα πρέπει να αναλάβουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν καλές επαφές, καλές διαδικασίες, υπάρχει το πρόβλημα του κατακαιρματισμού. Όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να θίξω εγώ είναι το θέμα της περιαγωγής. Είναι πάρα πολύ ακριβό, όπως ξέρετε, να χρησιμοποιήσει κανείς το κινητό του τηλέφωνο έτσι ώστε να κάνει κάποιες κινήσεις ε, ενώ ταξιδεύει στην Ευρώπη μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν τα προβλήματα των, των ανώτατων ορίων 3.000 ευρώ, 1.000 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σαφώς να το ρυθμίσουμε σαν εσωτερική αγορά. Οι τηλεπικοινωνίες και οι φορείς δεν ε, εκμεταλλεύονται αυτές τις δυνατότητες καθότι πλέον οι περισσότεροι αρνούνται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες καθότι είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Άρα υπάρχουν ευκαιρίες για τους φορείς τηλεπικοινωνιών, για τους οργανισμούς που μένουν ανεκμετάλλευτες και που θα μπορούσαν να αποφέρουν κάποια έσοδα αν ήταν λιγότερο ακριβά αυτές οι υπηρεσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πάλι αυτά τα νότα όρια 1000 ευρώ ανά γίγαμπάιτ παραδείγματος αν αυτή είναι η μία ε, λογική κατά την άποψή μου πρόταση Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για τους φορείς τηλεπικοινωνιών, αλλά αν δεν βρεθεί λύση, θα πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι χάνονται ευκαιρίες, ότι η κίνηση που θα μπορούσε να υπάρξει σε αυτή την ιστορική αγορά δεν ε, χρησιμοποιείται και μένουν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες και υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πέρσι έγινε μεγάλη εργασία από το Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν ήταν ε, αυτό που περιμέναμε όσον αφορά τις τιμές. Η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί όσον αφορά τον τομέα αυτό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το νέο φάσμα. Σαφώς και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Σήμερα δεν υπάρχει αρκετό φάσμα για την περιαγωγή των δεδομένων. Αυτή είναι η τεχνική, αν θέλετε, ε, δικαιολογία που μας δίνουν. Θα ήθελα κι εγώ, σαν σκιώδης ηγητής, να πω δύο λόγια. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Γενική Διεύθυνση της Εσωτερικής Αγοράς, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι επιτέλους μπαίνουμε στην ουσία, στα σοβαρά θέματα που αφορούν αυτήν την αγορά. Και μου φαίνεται ότι εδώ η Επιτροπή μας και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει ο εισηγητής, ο κύριος Αρίας, να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή αυτή έχει πραγματικές αρμοδιότητες όσον αφορά το θέμα αυτό και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. έχω ανησυχήσει κοιτώντα τα διάφορα σχέδια και τους τίτλους που δίνουν η μεν και η δε. Ψηφιακή αγορά. Μα πραγματικά ο ρόλος μας εδώ είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτής της έκθεσης. Τα βασικά εργαλεία που διαθέτουμε δεν είναι καινούρια. Είναι παλιά και τα έχουμε συζητήσει και ξανασυζητήσει εδώ σε αυτή την Επιτροπή εδώ και χρόνια στην οδηγία Η υπηρεσία παραδείγματο χάρη όσον αφορά τις υπηρεσίες παραδείγματος χάρη. Η υπηρεσία παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά και άλλες υπηρεσίες που εμπεριέχονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες δημιουργούν σήμερα προβλήματα και πιστεύω ότι ακούσαμε όλοι τον Ισπανό Υπουργό ο οποίος ήταν σαφέστατος για τα θέματα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν εμπόδια. Η Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2009 έπρεπε να υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την οδηγία αυτή. Δεν νομίζω ότι είδαμε τίποτα τέτοιο. Και όσον αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, σημειώνω ότι η Επιτροπή θα έπρεπε πριν το τέλος του 2009 επίσης να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές και για το θέμα αυτό. Δεν άκουσα τίποτα και δεν είδα τίποτα. Ίσως ε, πολύ σύντομα να το έχουμε. Έχω όμως την εντύπωση πραγματικά ότι όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά σημεία τα οποία συζητήσαμε είναι θέματα για τα οποία έχουν κατά καιρού συζητηθεί και προετοιμαστεί προτάσεις και νομοθετικά κείμενα, τα οποία όμως δεν βρίσκονται ολοκληρωμένα πουθενά. Παραδείγματος χάρη, το βαθμολόγιο των καταναλωτών, το θέμα της πολιτικής του ανταγωνισμού, το θέμα των δικτύων διανομής, πολλά προβλήματα που αφορούν τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν φτηνότερα προϊόντα μέσω του διαδικτύου, ακριβώς επειδή υπάρχουν οι περιορισμοί αυτοί τους οποίους γνωρίζουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε συνδυασμένα από κοινού και όσον αφορά αυτό το βαθμολόγιο θα πρέπει να ενσωματωθεί και αυτό το ζητήσαμε ήδη σε μια έκθεσή μας και το θέμα των ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών. Πιστεύω ότι το σύστημα πληρωμών, τα τεχνικά προβλήματα και εμπόδια και τα θέματα που αφορούν τους λογαριασμούς θα πρέπει να ειδωθούν από κοινά. Και δεν είναι διαφορετικό το ηλεκτρονικό εμπόριο από το παραδοσιακό εμπόριο. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, για τεχνικές, αν θέλετε, λύσεις, για την ίδια ακριβώς δραστηριότητα. Ο ρόλος μας λοιπόν εδώ θα πρέπει πραγματικά να ενισχυθεί κατά την άποψή μου. Δεν είναι θέμα ψηφιακό δεν πρόκειται για κάτι που αφορά αποκλειστικά και μόνο την φτηνή περιαγωγή δεδομένων, αλλά αφορά ένα θέμα το οποίο πρέπει να το απομυθοποιήσουμε γιατί ουσιαστικά αν βγάλουμε, αν θέλετε, την έγλη του διαδικτύου, πρόκειται για ένα απλούστατο θέμα βελτίωσης των διαδικασιών στην εσωτερική αγορά. Αφορά συναλλαγές της εσωτερικής αγοράς. Οι καταναλωτές, οι ευρωπαίοι καταναλωτές ουσιαστικά θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν τιμές και προϊόντα και να επιλέξουν πού θα αγοράσουν. Αν θα αγοράσουν σε μία, από μία αποθήκη που βρίσκεται στη δική τους χώρα ή κάπου αλλού στην Ευρώπη και ουσιαστικά όλες αυτές οι συναλλαγές τους επιτρέπουν καλύτερη, αν θέλετε, δυνατότητα επιλογής. Και όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε αυτό ακριβώς αφορούν. Οι εξαποστάσεως, εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ουσιαστικά διαφέρουν από το παραδοσιακό εμπόριο σε τομείς που δεν είναι ουσιαστικοί. Θα ξαναγίνω λοιπόν πρόεδρος, θα σταματήσω να είμαι σκιώδης εισηγητής και αφού ακούσουμε την Επιτροπή θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Ο Ντέιβιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις πολύ σημαντικές σας προτάσεις. Όσον αφορά το τελευταίο που είπατε, έχετε δίκιο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ουσιαστικά φαίνεται ότι αφορά καμιά φορά μόνο κάποιους ειδικού ή κάποιους ε, ε, οι οποίοι προσπαθούν ενώ ζουν σε μια ξένη χώρα να αγοράσουν προϊόντα από την πατρίδα τους. Είναι πολύ πιο γενικό το θέμα. Αν ένας καταναλωτής μπορεί να δει ένα προϊόν στο διαδίκτυο, να δει τις τιμές αυτό του επιτρέπει να πάει στο μαγαζί δίπλα στο σπίτι του και να διαπραγματευτεί καλύτερα το προϊόν που θέλει να αγοράσει σε ένα μαγαζί. Και ακριβώς αυτό πρέπει να προσφέρουμε σαν δυνατότητα στους καταναλωτές. Να συγκρίνουν, να δουν στο διαδίκτυο το τι συμβαίνει και ποιες τιμές προσφέρονται. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να βελτιωθούν οι εμπορικές συναλλαγές οι άμεσες Χρειάζεται λοιπόν κάποιοι καταναλωτές να γνωρίσουν τι τιμές προσφέρονται παντού στην Ευρώπη, να συγκρίνουν, να συγκρίνουν την ποιότητα των προϊόντων και κατόπιν να επηρεάσουν, γιατί περί αυτού πρόκειται, τις εμπορικές συναλλαγές οι τιμές online και offline, δηλαδή στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, θα πρέπει να είναι σχετικά συγκρίσιμες και κοντά. Και πιστεύω ότι ένα μαγαζί από τη στιγμή που θα ακούσει από πολλούς πελάτες του ότι οι τιμές του σε σύγκριση με αυτό που προσφέρεται στο διαδίκτυο είναι πολύ υψηλές, θα αλλάξει συμπεριφορά. Γιατί όταν μπαίνω σε ένα μαγαζί και βλέπω κάποιες τιμές που δεν ανταποκρίνονται στις τιμές που προσφέρει κάπου αλλού το διαδίκτυο, από τη στιγμή που αυτό θα γίνει ευρέως γνωστό, θα επηρεάσει και το λιανικό εμπόριο, το άμεσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν πολλά εμπόρια, εμπόδια. Υπάρχει το θέμα της έλλειψης εμπιστοσύνης, ένα τεράστιο πρόβλημα και το πρόβλημα των διαφορετικών κανονισμών και ρυθμίσεων. Αν κοιτάξει κανείς λοιπόν αυτές οι διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, διαπιστώνει ότι ο καταναλωτής θέλει να αγοράσει κάπου αλλού, προσπαθεί, υπάρχουν πάνω από 13,5 εκατομμύρια προσπάθειες, απόπειρες αγορών σε μια άλλη χώρα και τις περισσότερες φορές οι εταιρείε αρνούνται είτε να πωλήσουν είτε να στείλουν το προϊόν σε μια άλλη χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι η εμπιστοσύνη αυτή αυτή τη στιγμή είναι ελλειπής. Σιγά σιγά βελτιώνεται. Ακόμα και στο εσωτερικό μιας χώρας βλέπουμε ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξάνονται και βλέποντας τα αποτελέσματα των μελετών, τις απόπειρες που κάνουν οι Ευρωπαίοι να αγοράσουν κάποιο προϊόν σε μια άλλη χώρα στην Ευρώπη μέσω του διαδικτύου, αυτό μας δείχνει ότι η κατάσταση σίγουρα θα αλλάξει. Σήμερα βεβαίως βλέπουμε ότι υπάρχουν εμεί στα μεγάλα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη, των οποίων οι δυνατότητες να αγοράσουν στην ίδια τη χώρα είναι τεράστιες. Αν κάποιος όμως προέρχεται από την Κύπρο, παραδείγματο χάρη, οι δυνατότητες αποστολής των προϊόντων είναι ελάχιστες. Βλέπετε λοιπόν ότι οι δυνατότητες των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε τέτοιες μικρές ή απομακρυσμένες χώρες θα αυξηθούν πάρα πολύ εάν βελτιωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι περιφερειακές χώρες, οι μικρές χώρες θα πρέπει λοιπόν να επωφεληθούν από τη βελτίωση αυτού του εμπορικού δικτύου. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι χώρες παραδείγματος χάρη όπως το Βέλγιο που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης αντιμετωπίζουν κάποια τέτοια προβλήματα απομόνωσης γιατί χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, οι γειτονικές μεγάλες χώρες αρνούνται να τους ε, ε, τροφοδοτήσουν με προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη και θέμα συμπεριφοράς που πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο τελικά στον εισηγητή μας, τον κύριο Αρίας. Και θα ήθελα απλώς πριν του δώσω το λόγο να πω ότι από ό,τι βλέπω 7 Απριλίου θα υπάρχει μετάφραση της έκθεσης. 27 και 28 Απριλίου θα συνεδριάσουμε. 5 Μαΐου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τον Ιούνιο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί Ιούλιο ή Σεπτέμβριο. Το χρονοδιάγραμμα σας φαίνεται σωστό. Ευχαριστώ. Απλώς να σας πω ότι στις 7 Απριλίου εγώ πρέπει να δώσω την εργασία μου προς μετάφραση. Συνήθως ε, ε, παίρνει 10 μέρες περίπου η μετάφραση. Επομένως το νωρίτερο, 17 Απριλίου θα είναι έτοιμο το έγγραφο, διαθέσιμο δηλαδή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβαίνοντας και βεβαίως και κυρίως τους ε, σκιώδεις ε, ε, εισηγητές Νομίζω ότι η γενική κεντρική ιδέα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ίδια σε όλους μας. Ξέρουμε ότι και συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αρθούν και να έχουμε όλη κοινή θέση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, ε, υπάρχει μία λέξη την οποία σημείωσα σε όλες ε, τις παρεμβάσεις και που είναι πραγματικά η λέξη κλειδί, είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Μόνο με εμπιστοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά για να υπάρξει εμπιστοσύνη ε, θα πρέπει να υπάρξει απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά τα δικαιώματα τα οποία ήδη υπάρχουν και είναι θεσμοθετημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης ε, και τα, τις αρχές που ήδη διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και αφορούν την προστασία και των επιχειρήσεων και των ε, αγοραστών καταναλωτών. Βεβαίως να σας πω επίσης ότι είμαι απολύτως ερεθιμένος να ακούσω όλες τις προτάσεις εντός και εκτός της Επιτροπής ε, αν έχετε οποιαδήποτε πληροφόρηση βεβαίως να μου τη δώσετε και φυσικά θα συναντηθούμε, θα ήθελα να συναντηθούμε όσο γίνεται περισσότερες φορές με τους κοιότητες συγητής έτσι ώστε η εργασία να γίνει όσο ε, πιο πλήρης γίνεται. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την ε, Επιτροπή που μου έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ε, δεν απαντήσατε, ε, κύριε εκπρόσωπο της Επιτροπής, σχετικά με τον κατάλογο των ε, μη ικανοποιητικών πρακτικών. Έχει ολοκληρωθεί, ναι, ναι, έχει ολοκληρωθεί, τότε μπορείτε να μας τον στείλετε. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. με ενδιαφέρον παρακολούθησε αυτή τη συζήτηση η οποία κατέδειξε ότι όλοι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την, ε, ε, ενιαία, την εσωτερική αγορά, ε, όχι να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Παύλο Αρία Ετσεβερία και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Είναι η γνωμοδότηση του κ. Έγκστρομ, που νομίζω είναι η πρώτη γνωμοδότησή του στο Κοινοβούλιο. Είστε πρώτη φορά εισηγητή σε αυτή τη νέα θητεία. Επί της ουσίας ε, η υπεύθυνη είναι η βιομηχανίας νομίζω, η Επιτροπή Βιομηχανίας ε, και η ίντα έχει επίσης γνωμοδότηση. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Έγκστρομ για το ίντερνετ των πραγμάτων.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 θα μιλήσει κάποιο για, το, για τους εξονόμητους των Ο κύριος Μάντερ είναι εδώ. Ο κύριος ε, Νίκ. Ε, φαίνεται ότι δεν έχουμε πολλούς ε, σκιώδει Καλά, θα πάρω τη θέση του εάν δεν εμφανιστεί. Φαντάζομαι ότι ο καθηγητής κ. Κάμπος μπορεί ωραιότατα να μιλήσει εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Έγκστορμ, έχετε το λόγο. The way, the way I see the, uh, the, communication from, Η ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρούμε ότι είναι σημαντική και δεν έχει ιδιαίτερο νομοθετικό χαρακτήρα. Και εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω να υπάρχουν έτσι πολλά σημεία αντιπαράθεσης. Ίσως γι αυτό, εξηγεί και την απουσία των ε, σκιωδών εισηγητών. Συζητήθηκε σε πρώτη φάση το θέμα αυτό σε μια συνεδρίαση με περισσότερους, ε, περισσότερες παρουσίες. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση της Επιτροπής με μεγάλη σημασία για την Επιτροπή, τη δική μας. Καταρχήν ότι έχει σχέση με την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών. Εάν ξεκινήσουμε με συστήματα τα οποία κρατούν ίχνη από τα πάντα, παραδείγματο χάρη, από τη στιγμή που κάποιος θέλει να αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, αυτό γίνεται προσωπικό δεδομένο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι η κατηγορία και ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να επανεξεταστεί. Επίσης, και κάτι άλλο με το οποίο δεν συμφωνώ, το θέμα των προτύπων. Καταρχήν από την άποψη των ε, καταναλωτών αλλά ακόμα πιο σημαντικό μου φαίνεται για την εσωτερική αγορά κυρίως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εάν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές σε αυτό το νέο περιβάλλον θα πρέπει τα πρότυπα να είναι σαφή και για μια μεγάλη εταιρεία παραδείγματος χάρη τα ποσά που πρέπει να πληρώσουν παραδείγματος χάρη για να έχουν πρόσβαση σε αυτή την αγορά δεν είναι πρόβλημα. Για μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να είναι απαγορευτικά. Το διαδίκτυο λοιπόν ξέρετε ότι δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν κράτη-μέλη παραδείγματος χάρη που θεωρούν ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση στο ίντερνετ για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών που ενδεχομένως έχουν παραβιάσει κάποιους κανόνες. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ίση πρόσβαση. Αυτά προς το παρόν. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την ε, Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο τώρα στην σκιώδη συγκήτρια, την κυρία Κόμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όσα είπε, αυτά που είπε ο εισηγητής ε, καλύπτουν ε, την δυναμική και τα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά στο θέμα αυτό. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το υψηλό κόστος σύνδεσης δεν δίνουν ε, στην εσωτερική αγορά την ε, την δυνατότητα ε, αυτού της χρήσης του Internet of Things. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, το κυριότερο πρόβλημα πάντως το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι αυτό το οποίο σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών στοιχείων. Αυτή η προστασία της privacy λοιπόν είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Πρόεδρος, θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο εξ ονόματος των μη παρόντων σκιωδών εισηγητών τους φιλελεύθερους. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. E Εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ. Μιλήσατε για τις προκλήσεις, τις προηγούμενες οδηγίες οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν προκλήσεις για εμάς. Σαφώς και το θέμα του κόστους και της πρόσβασης είναι καθοριστικά. Και εγώ, επειδή ακριβώς δεν είμαι αρμόδια για το θέμα αυτό, θα ήθελα να πω γενικά ότι το θέμα του κόστους σαφώς και θα πρέπει να εξεταστεί στην ε, έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και προηγουμένως μιλήσαμε για τα δεδομένα, για τις πληροφορίες, για όλες αυτές τις ε, ροές ε, δεδομένων και πληροφοριών και το πιο σημαντικό είναι να βρεθούν μηχανισμοί οι οποίοι να βελτιώνουν τις διαδικασίες, οι οποίες να δίνουν περισσότερες πληροφορίες στον καταναλωτή. Μιλήσαμε επίσης εχθές και για το θέμα της σήμανσης και ο κύριος Μάντες ακριβώς έφερε εδώ ένα γυναικείο ένδυμα, ένα εσώρουχο αν θυμάστε, το οποίο ήταν εξαιρετικά μικρό, το οποίο όμως είχε δύο-τρεις τεράστιες ετικέτες με πάρα πολλές πληροφορίες επάνω ε, για να δείξει το παράδοξο κάποιες φορές των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Πολλές φορές όμως έχουμε πληροφορίες για προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα ή άλλα, άλλες ηλεκτρικές συσκευές περίπλοκες που σαφώς και χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ενημέρωση. Αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές πληροφορίες είναι απαραίτητες. Όπως επίσης εάν υπάρχουν ε, προβλήματα στα προϊόντα κατασκευής. Θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει ενημέρωση κατευθείαν στον καταναλωτή και εκ των υστέρων διόρθωση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ενσωματώσουμε. Επίσης, η ασφάλεια των δικτύων, κάτι που σαφώς και θα συμβάλλει στην καλύτερη και περισσότερη εμπιστοσύνη θέματα εσωτερικής αγοράς συμφωνώ μαζί σας. Θέματα που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Όσον αφορά τις συνοριακές εμπορικές συναλλαγές, οι κατασκευαστές των προϊόντων που στέλνουν τα προϊόντα σε μια άλλη χώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες που παρέχονται στο διαδίκτυο. Και ξέρουμε ότι η επίδραση των πληροφοριών που υπάρχουν ε, στο διαδίκτυο για παραδείγματο χάρη φτηνά προϊόντα σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρονται στο διπλανό μαγαζί σίγουρα είναι κάτι που με τον καιρό θα έχει κάποιες επιπτώσεις στην τοπική αγορά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν κύριε Έγκστρομ για τις προτάσεις σας. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή τον κύριο Ματέο Γκόγια Μανουέλ. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, σύντομη και πλήρη παρουσίασή σας. Συμφωνούμε με αυτά που είπατε. Και... Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι οι οποίοι τοποθετήθηκαν συμφωνούν. Και δεν έχω και πολλά να σας προσθέσω. Απλώς θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, ότι ε, εκτός από όλα τα άλλα τα οποία προτείνουμε, έχουμε και αυτόν τον ε, διοργανικό διάλογο, Οπότε γι' αυτό και είναι πολύ θετικό ότι τα λέμε τώρα εδώ και σε άλλες κοινωνικές επιτροπές γιατί αυτό ακριβώς είναι στο πνεύμα που διαπνέει και τη δική δράση. Και τώρα κάτι άλλο σημαντικό το οποίο έχει να κάνει με τα, τα, τα πρότυπα αυτά, γιατί δεν είναι δυνατόν το ένα θέμα να θεωρηθεί άσχετα από το άλλο. Έχουμε την πρώτη γραμμή δράση που αφορά την ε, ανακοίνωση και είναι αυτή η διακυβέρνηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ούτε είναι δυνατόν να το αποσυνδέσουμε το θέμα των, ε, ε, των προτύπων γιατί το ένα θέμα λειτουργεί υπό την προπόθεση του άλλου και άρα ε, είναι πάρα πολύ θετικό το πώς ε, προσφέρετε και εσείς τις απόψεις σας τα βλέπετε επίσης για την προστασία των δεδομένων νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί μια συνένεση μεταξύ ημών ε, και ημών γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα πρέπει στην ανακοίνωση να αφιερώνουμε αρκετό κείμενο σε αυτό το θέμα και γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το ζήτημα όπως ακριβώς ξεκινήσαμε με την σύσταση η οποία τον Μάιο πέρυσι ε, εγκρίθηκε για την προστασία του ιδιωτικού βίου και των σχετικών δεδομένων. Για να ολοκληρώσουμε τώρα ένα πραγματάκι ακόμα που θα πρέπει να σας τονίσω είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο. Πρόκειται για αυτή την διάκριση που θα πρέπει να γίνει μεταξύ το, του, του ενός ίντερνετ και, και του, του άλλου, του υπολείπου ίντερνετ, γιατί το, το, το, ένα, το ένα είδος ίντερνετ ε, αφορά την Ευρώπη, αφορά την, ε, την ε, βιομηχανία, ε, και αφορά και τους διεθνείς μας εταίρους. Όμως αυτό απλώς είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία, μία σαν τις άλλες, το ίντερνετ των πραγμάτων. Και το αναφέρει γι' αυτό και ανακοίνωση κάνει αυτή την ημερομηνία, παραπέμπει στις διάφορες τεχνολογίες. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε αυτή την διάκριση και θα πρέπει άρα να προσέξουμε και την διατύπωση. Τώρα, δεν μπορώ να υπησέλθω στις λεπτομέρειες, αλλά αν έχετε κάποιες ε, ε, ερωτήσεις, ευχαρίστως να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε την Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Και σε λίγο θα δευτερολογήσει ο κύριος Άγκστρομ. Αλλά, για να δούμε, τι χρονοδιάγραμμα προβλέπετε. Και πέστε μας, εάν συμφωνείτε. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Τρίτου, το μεσημέρι. 7 και 8 θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε. 4 Μαΐου θα γίνει η ψήφιση, άρα θα πρέπει να προσέξουμε. Κύριε Ισηγητά, έχετε κάτι να αναφέρετε για να ολοκληρώσουμε. Όχι, δεν έχω και πολλά να σας πω. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέσχουν. Κανένα πρόβλημα και με το χρονοδιάγραμμα. Άρα όλα καλά. Πολύ χαίρομαι που είστε ικανοποιημένος, λέει ο πρόεδρος. Επίσης, πάμε τώρα στο τελευταίο μας θα είναι τελευταία έκθεση για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Συνεχίζουμε με τα ζητήματα τα οποία αφαιρούν το διαδίκτυο και την οικονομία. Αφορά την διακυβέρνηση του ίντερνετ. Τα επόμενα βήματα. Η κυρία Νίμπλε είναι εδώ. Η κυρία Σουλιέ ε, που έχουν επεξεργαστεί το θέμα πολύ καιρό. Ποιος θα μιλήσει από την Επιτροπή. Κυρία Νίμπλου. Ο κύριος Μάρκο. Μπορείτε και οι δύο να δείτε το λόγο γιατί έχουμε το χρόνο, λέει ο πρόεδρος. Πολύ χαίρομαι που η κυρία Στάιλς πρόκειται επίσης να... Στάιλ, Στάιλ, να, να, να μας πει ε, για την δική της γνωμοδότηση. Και εγώ έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα της. Είμαι και σκιώδης. Άλλο σκιώδης. Για την ΚΟΕ ποιος είναι, κύριος Άγκστρομ, εσείς είστε ο σκιώδης για την ΚΟΕ. Γιατί νομίζω ότι έχετε τα, τα προσόντα. Οπότε να σας κάνουμε εμείς σκιώδη. Οι φιλελεύθεροι. Οι φιλελεύθεροι ερημοδικούν σε καθηγητή Κάμπο, ε, βλέπω κόσμο εδώ που θα μπορούσε να συμβάλλει. Οπότε, κυρία Στάιλερ, μπορείτε να λάβετε το λόγο και να παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του συναδέλφου. Ξέρετε, ο παλιό Κιώδης ήταν ο κύριο Μπαρνιέ. Και χθε τα είπαμε τον τωρινό αντικαταστάτη του. Πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ χρήσιμα είναι τα όσα είπαμε και οπότε αν έρθει θα είναι ακόμα καλύτερα. Όλα εδώ για αυτή την έκθεση ξεκινούν από ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα το οποίο ονομάζεται διακυβέρνηση του ίντερνετ τα επόμενα βήματα. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί ποιος θα σκεφτόταν ότι κάτι το οποίο θεωρήθηκε πολυτέλεια θα καταλήξει μια αναγκαιότητα, κάτι απαραίτητο στην διεθνή ζωή. Είδατε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και αν ρίξει κανείς μια ματιά στον αρχό της Επιτροπής θα διαπιστώσει ότι πάρα πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ίντερνετ. Τα αναφέρει η Κομισιόν και έχουμε και αυτή την IETF, αυτή την Task Force των Μηχανικών. Μιλούμε για ε, μη κυβερνητικό όργανο, ομάδα και άρα θέλουμε να δούμε εδώ πέρα πώς θα είναι δυνατόν να πανεύει κανείς όταν κάτι πάει στραβά σε σχέση με το ίντερνετ. Ε, να, ε, λοιπόν, ένα, ένα θεματάκι. Αλλά έχουμε και άλλους δύο φορείς που δεν βλέπω ότι πρέπει να σας αναφέρω και είναι το Internet Assigned Numbers Authority. IANA. Και άλλο ένα που αφορά τα ονόματα και τους αριθμούς, ε, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό από διακυβέρνηση που επίσης ε, είναι σημαντικό, είναι και αυτή η μη κερδοσκοπική οργάνωση, είναι σωματείο. Και ξέρετε, ε, όλοι αυτοί θα συναντηθούν, θα συναντιόνται συνέχεια στις Βρυξέλλες. Να γιατί αυτό έχει πάρα πολύ σημασία για το κείμενό μου. Για ρίχτε μια ματιά τώρα στα της διακυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε ποιε είναι οι αρχέ που διαπνούν τη διακυβέρνηση του, του Ιντερνετ. Ε, ε, να υπάρχει διαλειτουργικότητα, να υπάρχει μια τέτοια αρχιτεκτονική η οποία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και ε, θα πρέπει άρα η διαχείριση που γίνεται σήμερα να μην έχει διακοπή, να λάβουμε υπόψη τους διάφορους πόρους του παγκόσμια σε παγκόσμια, παγκόσμια ισχύ ε, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στο Ιντερνετ ε, και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς θα γίνει αυτή η διακυβέρνηση. Όμως τελικά το σημαντικό είναι να δούμε στο μέλλον, στα επόμενα 10-20 χρόνια, τι εξελίξεις θα έχουμε, ποιες θα είναι οι προκλήσεις και τι μπορούμε από κοινού να κάνουμε θα πρέπει να υπάρχει διακυβερνητικός διάλογος. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια ε, αντιμετώπιση. Και εδώ λέμε για υποχρέωση λογοδοσίας, μιλάμε για διαφάνεια, όλα αυτά είναι σημαντικά. Όλα αυτά θα πρέπει να διεκπεριωθούν και έτσι να μπορέσουμε κάπου να καταλήξουμε Έχουμε επτά σημεία, επτά παραγράφους σε αυτό το κείμενο, ό,τι θεωρώ πιο σημαντικό. Και τα βασικά είναι τα εξής. Ότι εντείνεται η χρήση από καταναλωτές, εταιρείε και αρχές. Οπότε έχουμε την περαιτέρω ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς. Θα τα συζητήσαμε και χθε. Και είναι πάρα πολύ προβεβλημένο το Ιντερνετ για κοινωνικές, για εμπορικές δραστηριότητε, χρειάζεται συντονισμό περισσότερος. Θα πρέπει αυτό να θεωρηθεί ότι είναι δημόσιο συμφέρον. Και ε, καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητεί σε αιτήσια βάση με τους εμπλεκόμενους. Τα είπε και χτες η σχιώδη Ιδρύα του ΕΛΚ. Γιατί να μην τα συζητούμε και εμείς σε θεσμική βάση κάθε χρόνο. Και ε, είπαμε, η ICAN, αυτός ο, ο φορέας, ε, πρόκειται να συναντηθεί στις Βρυξέλλες. Εμπόριο, πληροφορίες, ονόματα, ε, είναι αυτή η υπηρεσία πάρα πολύ σημαντική. Και επίση έχουμε και μια γνωμοδότηση τη Επιτροπή Πολιτισμού πάνω σε αυτό, γιατί χρειάζεται τελικά να λάβουμε υπόψη το ποια είναι η κυρία αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Βιομηχανία, γιατί είναι και θέμα τη προστασία των ανηλίκων. Και αυτό είναι η διακυβέρνηση του Ιντερνετ. Ε, επίσης ζητούμε οι εμπλεκόμενες εταιρείε να διευκολύνουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και τι σχετικές συναλλαγές. Να είναι προσβάσιμη αγορά και στους ε, νέους που μπορούν να μπουν στον παιχνίδι του ανταγωνισμού. Βέβαια, έχουμε ακούσει ένα σωρό απόψεις και θα δείτε, υπάρχουν διάφοροι σκιώδει ηγητέ από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε. Όμω, συμπαθάτε μα γιατί τελικά δεν τα καταφέραμε να κάνουμε όλοι μαζί μια συνάντηση. Γιατί ήταν τόσο πολύ ο χρόνο που είχα για να κάτσω να γράψω το κείμενο και από την άλλη μεριά ούτε ξέραμε ποιο είναι ο σκιώδε από ποια πολιτική ομάδα. Γι' αυτό σα λέω ότι ό,τι μου είπαν είναι πάρα πολύ πολύτιμο και νομίζω η καταληκτική ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα τη τροπολογία την επόμενη εβδομάδα, έτσι δεν είναι. Οπότε και, τελικά γυράσκω ήδη διδασκόμενοι. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Στάιλερ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά τα θίξατε και ήδη όλα αυτά τα αρκτικόλεξα τα ξέρετε γίνεται αητός σε αυτά. Λοιπόν, όμως δεν βλέπω άλλον σκιώδη. Αλλά όποιος άλλο τυχόν θέλει να λάβει το λόγο αυτό, θα πρέπει να μιλήσει πρώτο, μια που είμαι πρόεδρο Κριστιαν. Να, ο, πιο φρέσκος από τους σιώδης συγκριτές. Μόλις τον Συμφωνώ με την όλα αυτά που είπατε, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί ακριβώς όπως είπατε και εσείς δεν είναι παιχνίδι το Ιντερνετ, είναι τμήμα της κοινωνίας. Ναι, μόνο είχαμε μια εβδομάδα, δεν, είχαμε, δεν θα έχουμε κανέναν εξπέρ. Αλλά για την ICAN ε, πρέπει κάτι να γίνει, κάποια επαφή να γίνει. όλα, ναι σε όλα, πρόεδρος. Α, να ήρθε μια ο ε, μισό λεπτό για να, να ξελαχανιάσετε, ε, επιταχύναμε πολύ, είμαι σίγουρος ότι θα σας σφυρίξουν το ότι συζητήσαμε και να σας πω από πλευρά της δικής μου πολιτικής ομάδας. Και μετά η συνάδελφος θα λάβει το λόγο. Εγώ ξέρετε ενδιαφέρομαι για το θέμα. Γιατί έχω πάει σε όλα τα φόρουμ για την διακυβέρνηση του ίντερνετ και είχαμε και τους ε, συναδέλφους της Κομισιόν που έχουν έρθει σήμερα εδώ, είναι πολύ δυναμική δραστήρια γιατί για την υπόθεση αυτή τη διακυβέρνηση έχει παίξει σημαντικό ρόλο η Κομισιόν. Στα σοβαρά έχει ασχοληθεί πολύ καιρό, οπότε. Είχαμε και επίσης τις συναντήσει κορυφή, τη παγκόσμια για την κοινωνική πληροφορία, συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Αλλά έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Χρειάζεται η σταθερότητα που νομίζω ότι θα επιφέρει η ICAN. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Για ένα πολύ σημαντικό θέμα παγκόσμιας εμβέλεια. Ο βασικός στόχος είναι να μην έχουν πολιτικοποίηση, και ειδοποιήσει. Θέλουμε να είναι ανοιχτό το Ιντερνετ, να μην υπάρχει κάτι που να μην είναι τόσο φιλικό στο χρήστη. Βέβαια υπάρχουν πολλέ απόψει, συμφωνούν όλοι σε όλα αυτά. Και είπαμε για τον κυβερνητικό έλεγχο τι μπορεί να γίνει. Ο ρόλος του Υπουργείου Εμπορίου γιατί οι αρχέ του Ιντερνετ ανάγονται στις ΗΠΑ, οπότε το δικό του Υπουργείο μπορεί, έχει σημασία το τι λέει, τι κάνει. Και μιλάμε για αυτή την εταιρική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Εμεί όμω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποια σταθερότητα, κάποια συνέχεια και να συμβάλλουν να εμπλέκονται αυτοί που θέλουν να προχωρήσει η υπόθεση και όπως μας είπε και η συγκήτρια έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία αποτελούν ένα καινούριο κόσμο και είναι απλώς αφετηρία τους η υπόθεση της διακυβέρνησης. Ας πούμε τα τεχνικά πρότυπα. Ήδη έχουμε κάνει ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα τεχνικά πρότυπα. Έχουμε και έκθεση που αφορά τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία όμως εξελίχθηκαν για το Ιντερνετ. Και είναι θέμα κάποιων μηχανικών, κάποιων ειδικών που πρέπει να εξασφαλίσουν την εύρετη λειτουργία του διαδικτύου. Και ήρθε στη συνάντηση κορυφής ο ίδιος, ο εμπνευστής, ο εφευρέτης του διαδικτύου, του παγκόσμιου ήρθε να μας μιλήσει. Και ε, χάρη σε αυτόν έχουμε αυτή την τρομερή δυνατότητα το να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε τόσα πράγματα λόγω της εξέλιξης του λογισμικού του λογισμικού ιδίως ανοιχτής πηγής επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να ε, περιφρουρηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως είπε η κυρία Στάιλερ Επίσης, ο, ο έλεγχος των ονομάτων που έχουν εμπορική αξία. Domain names. Είναι κάτι σαν εμπορικά σήματα. Και έχουμε το cyber squatting, όπου κάποιοι κατοχυρώνουν κάποια σήματα και κατόπιν τα πουλάνε στον, σε αυτόν που θεμητά τα χρησιμοποιούσε αρχικά. Άρα, Χρειάζεται η διακυβέρνηση να παρέμβει εδώ. Πέρσι όμως αυτά συζητήθηκαν. Ήμουν και εγώ και εκεί και άλλοι συνάδελφοι στην άντληση της ΆΙΚΑΝ, την περσινή. Κάθε συνάντηση της ΆΙΚΑΝ αξίζει να πάει κανείς και μπορεί γιατί αυτές είναι δημόσιες. Οπότε είχαν ε, βάλει μια πλατφόρμα με ένα τραπέζι με στη μέση, γύρω γύρω ήταν το κοινό και τους άκουγε, τους έβλεπε. Αλλά πάρα πολύ βασικό ήταν το ότι αποφασίστηκε να να απελευθερωθούν δύο καινούρια ε, αρχικά που κολλάνε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ας πούμε το, όπως το EU. Και αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια τεράστια ποικιλία χώρων γιατί βέβαια είναι επιπερασμένος ο αριθμός των ε, domain names αυτών των αρχικών τα οποία διατίθενται. Ένα σωρό θέματα έχει καλύψει η κυρία Στάιλερ. Επιδέχονται αυτό και κάποιες συμπληρώσεις. Αλλά νομίζω ότι μια που είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα θα πρέπει η Επιτροπή μας κάτι να φτιάξει. Τώρα, ξαναφοράω το καπέλο του Προέδρου και δίνω το λόγο στην συνάδελφο που είναι καινούριο μέλος. Καλώς ορίσατε και έχετε το λόγο σαν σκιώδη συγκεκριμένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησα. Ζητώ συγγνώμη από εσάς από τον εισηγητή, τον οποίο δεν μπόρεσα να ακούσω, και από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Διαπιστώνω ακούγοντάς σας ότι δεν είναι εύκολο να μπορεί κανείς να είναι παρόν σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ λοιπόν καταρχήν που μου δίνετε το λόγο και θα ήθελα να πω ότι η πρόταση αυτή της Επιτροπής είναι πλήρης, είναι σε γενικές γραμμές επικοδομητική και επιμένει ιδιαίτερα στον κεντρικό ρόλο που μπορεί να παίξει εδώ ο ιδιωτικός τομέας στη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Πιστεύω ότι θα πρέπει και εμείς στη γνωμοδότησή μας να υπογραμμίσουμε αυτό το ρόλο, να τον ενισχύσουμε. Το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κανέναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης που προσφέρει ίσες εγγυήσει όπως ε, αυτή τη στιγμή αυτές που προσφέρονται από τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να το υπογραμμίσουμε αυτό και παρόλα αυτά να πούμε ότι σαφώς και οι δημόσιες πολιτικές και οι πολιτικές κοινής ωφέλειας είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πρέπει να ξανασκεφτούμε το ρόλο αυτών των πολιτικών, να δούμε τι μηχανισμοί μπορεί να ακολουθηθούν εδώ από τους ιδιωτικούς φορείς που σήμερα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διακυβέρνηση του ίντερνετ έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και πιο υπεύθυνο τρόπος διακυβέρνησης. Διαφάνεια λοιπόν και αρμοδιότητες όσον αφορά την διακυβέρνηση. Δεν ξέρω τι είπαν ακριβώς οι προηγούμενοι ομιλητές, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε η πρόταση της Επιτροπής, υπεγράφει μια νέα συμφωνία μεταξύ του ICAN και του, της Αμερικανικής Αρχής. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό καθότι έτσι ξεκίνησε και η μεταρρύθμιση, η θεσμική μεταρρύθμιση του ICAN και για να παραμείνουμε απαιτητικοί όσον αφορά τη διαφάνεια ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε εδώ και κάποιες προτάσεις Όσον αφορά τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα από τις τέσσερις επιτροπές, τα τέσσερα πάνελ που ξεκίνησαν την εσωτερική αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση του ICAN. Υπάρχουν, όπως ξέρετε φαντάζομαι, τέσσερις φορείς ανεξάρτητοι, τέσσερα πάνελ ανεξάρτητα, τα οποία λειτουργούν ε, από το φθινόπωρο του 2009 και για να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, καλό θα ήταν κατά την άποψή μου να ζητήσουμε μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων εργασίας αυτών των ομάδων εργασίας ή πάνελ ή επιτροπών, όπως θέλετε ε, ονομάστε τα πάνελ, επαναλαμβάνω, που εργάζονται με ανεξάρτητο τρόπο στο εσωτερικό του ICAN. Αυτό θα μπορέσει να είναι πολύ χρήσιμο, πιστεύω, στη γνωμοδότηση του εισηγητή. Ίσως, επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των κυβερνήσεων. Επουδενή λόγο δεν θέλω να αμφισβητήσω τη σημερινή διακυβέρνηση του ίντερνετ. Τίποτα το επαναστατικό δεν θέλω να κάνω εδώ, αλλά επειδή πρέπει να λειτουργήσουμε σε διεθνές επίπεδο, σε πολυμερές επίπεδο και σε πολυεθνικό επίπεδο, ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε και το ρόλο των κρατών, των κρατικών αρχών στη διακυβέρνηση του διαδικτύου μέσω ίσως του φορέα του συνδετικού κρίκου που σήμερα λειτουργεί μεταξύ των κυβερνήσεων και του ΆΙΚΑΝ, της συμβουλευτικής αυτής ομάδας. Δεύτερος άξονας λοιπόν που θα πρέπει να εξεταστεί είναι ο τρόπος συνεργασίας, καλύτερης συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και ICAN πάντα σε μια πολυεθνική, πολυμερή ε, βάση και χωρίς να ανατρέψουμε τίποτα από αυτά που σήμερα λειτουργούν. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προτείνω είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το σημείο 4 της εισήγησης. Παρουσία ενός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επόμενη συνάντηση του ICAN στις Βρυξέλλες, τον Ιούνιο. Εγώ προσωπικά θα ήμουν σαφέστατα υπέρ. Θεωρώ ότι το ICAN βεβαίως και θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του με την παρουσία ενός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου που έχει ήδη συνεδριάσει αρκετές φορές επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει επίσης και σε αυτές τις συνεδριάσεις πιστεύω στο μέλλον να συνεδριάσει. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Βίλνιους πριν το τέλος του χρόνου. Η συμμετοχή μας σε αυτό το φόρουμ συντονισμού θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αυτά ήθελα να πω. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι που δεν έχει άμεση σχέση με το μηχανισμό διακυβέρνησης, αλλά να πω ότι ίσως αυτή η γνωμοδότηση που θα προετοιμάσουμε θα μπορούσε να συμπληρωθεί από μία αναφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Κάτι το αλληλένδετο με όλες τις αρχές που προωθούμε. Μιλήσατε για την ενίσχυση κατά τους εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και πιστεύω ότι και το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά σημαντική η πνευματική ιδιοκτησία και η προστασία της, αλλά και η σημασία του διαδικτύου για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, η καταπολέμηση των ε, πλαστών προϊόντων, της πειρατείας. Το διαδίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο για την καλύτερη οργάνωση, την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεν πρέπει όμως επειδή είναι λόγο να δημιουργήσουμε εδώ έναν χώρο στον οποίο όλες οι ανεξέλεγκτες και οι κλιματικές συμπεριφορές θα μπορούν να εκφραστούν. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία. Τη συγχαίρω γιατί πραγματικά είναι πολύ προσεκτική στις προτάσεις όλων. Την ευχαριστώ για την μέχρι τώρα εργασία της και την παρακαλώ να λάβει υπόψη της και αυτά που προτείνουν εδώ στην συνεδρίαση οι διάφοροι μιλητέ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και ο κύριος Ζουβέ θέλει να μιλήσει, νομίζω τον έχω στο κατάλογό μου. Α, και ο κύριος Μπουζόη. Ζητώ το λόγο ενώ δεν είμαι εισηγητής και ο εισηγητής είπατε ότι έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε μια άνεση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πάρω το λόγο να πω τρία πράγματα. Ε, να αναφερθώ λοιπόν στο ΙΚΑΝ. Σύμφωνα με αυτά που όλοι λένε και γράφουν, ε, το ΙΚΑΝ προφανώς εξελίσσεται προς τη κατεύθυνση και θα ήθελα να έχουμε ε, μια έκθεση όσον αφορά, έναν απολογισμό δηλαδή, όσον αφορά τις τελευταίες ε, εξελίξεις, ε, κυρίως σχετικά με την εξέλιξη των ιδιαίτερων σχέσεων μεταξύ του ΙΚΑΝ και της Αμερικανικής κυβέρνησης. Βεβαίως τα πράγματα εξελίσσονται, αλλά θέλω να, θα ήθελα να μάθω πού βρισκόμαστε. Δεύτερον, το δεύτερο σημείο ενδεχομένως ξεπερνάει λίγο το θέμα μας, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε και το ερώτημα αυτό. Το ίντερνετ βεβαίως είναι ένα εργαλείο δημοκρατίας. Η δημοκρατία στη διάρκεια ε, του ρου χρησιμοποίησε τις ε, τεχνολογικές εξελίξεις κάθε φορά, ξέροντας ότι Μερικές χώρες κλείνουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, απαγορεύουν το διαδίκτυο, την πρόσβαση στο διαδίκτυο ε, έτσι ώστε να εμποδίσουν την ελευθερία έκφρασης ε, και την συμμετοχή σε θέματα τα οποία μας φαίνονται απολύτως ε, ουσιώδη για την δημοκρατία. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα αυτό σήμερα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τις δυνατότητες, τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε την ελευθερία της πληροφόρησης σε όλες τις χώρες. γιατί τότε θα έχουμε παίξει τον ρόλο μας βεβαίως ε, ακόμα καλύτερα γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε κυρίως να ασχοληθούμε με την εσωτερική αγορά αλλά θέλουμε οπωσδήποτε και να παραμείνουν εν ζωή κάποιες σημαντικές γενικές αρχές. Τρίτο θέμα, πνευματική ιδιοκτησία και λυπάμαι που δεν εμφανίζεται πουθενά αυτή η λέξη στον κατάλογο των προτάσεων. Είναι και αυτό ένα από τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Γενετικού Κώδικα. Είναι στο γενετικό μας υλικό εγγεγραμμένο ε, αυτό το θέμα και επομένως μέσω της διακυβέρνησης του διαδικτύου πρέπει οπωσδήποτε να υπεραμεινθούμε και αυτού του στοιχείου και εν πάση περιπτώσει να σας, το πω, λίγο πιο διακριτικά, εάν εμφανιζόταν αυτή η έκφραση, η πνευματική ιδιοκτησία στο κείμενο, δεν θα μας κακοφαινόταν καθόλου. Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, ιδιαίτερος είναι προσφυλές στην Ευρώπη. Κύριε Μπουρζόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να καλωσορίσω την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν. Καθώς επίσης ε, και την γνωμοδότηση της κυρίας ε, Στάιλερ τα σημεία τα οποία έχουν υποβληθεί στην συζήτηση καλύπτουν νομίζω τον προβληματισμό μας όσον αφορά ε, την ανάπτυξη του, της διαδικτυακής αγοράς και την προστασία των, ε, αγορό, των ε, καταναλωτών. Νομίζω ότι κυρίως η καταπολέμηση ε, του κυβερνοεγκλήματος, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ε, γιατί όταν ε, αναφερόμαστε κυρίως σε στην προστασία των ανηλίκων καθώς επίσης και την προστασία των προσωπικών στοιχείων του καθενός μας τότε το θέμα αποκτά πολύ σημαντικές διαστάσεις. Επίσης, ε, θυμάμαι μακρές συζητήσεις ε, που είχαμε οποτεδήποτε χρειάστηκε να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα ε, στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον χώρο και από την άλλη πλευρά να διατηρήσουμε τον αστικό χαρακτήρα του διαδικτύου. Δεύτερο στοιχείο συζητούμε διαρκώς την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τον αυξανόμενο αριθμό ε, των διασυνοριακών online συναλλαγών. Λέμε λοιπόν ότι η βελτίωση των συνδικών πρόσβασης στο ίντερνετ θα έχει καλό θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή αγορά. και κατά αυτή την έννοια λέω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η ασφάλεια όλων αυτών των συναλλαγών. Εάν οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι βέβαιοι, έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα, είναι βέβαιοι ότι θα προστατευθούν τα προσωπικά τους δεδομένα τότε εάν ήταν βέβαιο ότι οι δικτυακές πύλες τις οποίες επισκέπτονται είναι ασφαλείς, τότε σίγουρα θα είχαν πολύ μεγαλύτερη βούληση να ε, ε, συμμετέχουν ε, στο διαδίκτυο και επομένως στο εμπόριο μέσω του διαδικτύου. Περαίνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά την εισηγήτρια και να την συγχαρώ. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες αλλά ελπίζω ότι κάπου θα τα βρούμε η συγγήτρια κι εγώ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Uh, Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να πει δύο λόγια, να σχολιάσει όλα αυτά που ακούστηκαν και ενδεχομένως να προσθέσει και κάποια επιπλέον στοιχεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σημείωσα την ισχυρή αναφορά όλων σε ορισμένα στοιχεία τα οποία ήδη περιέχονται στην ανακοίνωση. Ταυτοχρόνως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ρόλος, δημόσιος ρόλος για την διακυβέρνηση του ίντερνετ και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Η σταθερότητα, ας πούμε, δεν ιδιωτικοποιείται και ενδεχομένως ε, ε, κάποια εμπορική συναλλαγή θα αφορά ας πούμε το Λος Άντζελες αλλά παρόλα αυτά το κοινοβούλιο θα έρθει μετά και θα ρωτήσει τι κάνατε έτσι ώστε να είναι ασφαλής να προστατευτεί ο πολίτης ο οποίος έχει προχωρήσει σε αυτήν την ε, συναλλαγή. Ε, είναι γεγονός ότι, και το έχουμε πει άλλωστε, ότι αυτή η διακυβέρνηση ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είναι ένα μοναδικό ε, φαινόμενο κατά κάποιο τρόπο Βεβαίως εμείς εργαζόμαστε ε, όσον αφορά το μέλλον του εικόν ε, και με τις Ηνωμένε Πολιτείε δουλεύουμε πολύ στενά, συνεργαζόμαστε πολύ στενά έτσι ώστε να συμμετέχουμε στις ε, διαδικασίες αυτές. και πρέπει να πω ότι τώρα θα αρχίσει να εγκαθίσταται το πρώτο πάνελ They Αναθεώρησης. Είναι γεγονός ότι δυσκολευτήκαμε λίγο για να δούμε τι, με τι ακριβώς θα ασχοληθεί και ποιοι ακριβώς θα αποτελούν αυτό το review panel, αυτό το panel αναθεώρησης. Και ξέρετε βεβαίω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θα είναι στη διάθεσή σας έτσι ώστε να κάνει ένα απολογισμό και να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Ο ρόλο του Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, στο ζήτημα αυτό. Βεβαίως, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι σαφής και δυνατός, γιατί άλλωστε είναι δυνατή πάντα η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Και ε, πραγματικά σας διαβεβαιώνω ότι η αντιπροσωπεία και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέβασε το επίπεδο της ευρωπαϊκής ε, παρουσίας και γνωρίζουμε ότι και ο πρόεδρος ήταν μέλος της αντιπροσωπείας. Τώρα κάποια στοιχεία όσον αφορά κάποιες ε, προτάσεις που ακούστηκαν. Ε, αναφέρεστε σταθερότητα. Ναι, βεβαίως. Η σταθερότητα αποτέλεσε το κυρίαρχο στοιχείο, το διαρκώς επαναλαμβανόμενο στην διάσκεψη κορυφής για την ασφάλεια διαδικτύου και τη διακυβέρνηση, ε, του ε, διαδικτύου. Βεβαίως η σταθερότητα και η σταθερότητα της πληροφορίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, επίσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πιο υπόλογες. Ναι, φυσικά, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στην εθνική κυριαρχία ε, όσον αφορά ε, δικτυακούς τόπους όπως ας πούμε το .be, .gr ε, και το .com. Και ήδη ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα ανοίξει ένα μεγάλο κουτί στο ICOM, δηλαδή αυτά τα νέα GTLTs. Ενδεχομένως θα υπάρξουν νέες διευθύνσεις όπως τελεία Berlin. Εν πάση περιπτώσει εδώ είναι μια διαδικασία η οποία θα συζητηθεί και στις Βρυξέλλες. Αυτό με φέρνει στο θέμα της, της συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Και όπως είπατε και εσείς κυρία Στάιλερ, η συνεδρίαση αυτή ε, θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες. Είναι σαφές, σαφέστατο μάλιστα, ότι οι συνεδριάσεις αυτές είναι απολύτως ανοιχτές. Παραμένει βεβαίως μια συμβουλευτική επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι συνεδριάσεις ανοιχτές όπου ο καθένας μπορεί να είναι παρόν καθένας μπορεί να παρίσταται. Όσον αφορά το cyber το, το έγκλημα ε, ε, στον, ε, στον χώρο και όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να πω ότι στις συνεδριάσεις της εικόνα έχουμε πολύ αναφερθεί στο θέμα της εφαρμογής ε, των νόμων ε, και της ε, δίωξης οποιονδήποτε καταπατούν το νομικό πλαίσιο, οποιουσδήποτε παραβιάζουν το νομοθετικό πλαίσιο. Και επομένως ο χώρος αυτός, η κοινωνία αυτή δεν είναι μια περιοχή χωρίς νόμο Βεβαίως εφαρμόζεται η νομοθεσία για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικής ζωής. Αυτά ήθελα να πω. Αλλά κυρίως να ευχαριστήσω πραγματικά το Κοινοβούλιο γιατί έχει τόσο πολύ αναμειχθεί, τόσο ενεργά έχει αναμειχθεί σε αυτά τα θέματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που παίζεται τόσο πρωταρχικό ρόλο σαν κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και εμείς ε, ε, κύριε Νίμπο. Και είδα και εγώ τον τρόπο με τον οποίο ηγηθήκατε της ε, ICON και πραγματικά μου δώσετε και τη δυνατότητα να κατανοήσω καλύτερα κάποια θέματα τα οποία αγνοούσα. Κυρία Στάιλερ. «22 Μαρτίου τροπολογίες 7 Απριλίου συζήτηση, 8 Απριλίου ψηφοφορία. Συμφωνείτε? Θέλετε να πείτε και δύο λόγια ολοκληρώνοντας. Δύο λόγια μονάχα. Έχω την αίσθηση ότι μπορώ στην ε, προσπάθειά μου να ολοκληρώσω την εργασία μου ε, ενδεχομένως να δω και ε, την εργασία της ICAN μέχρι τώρα να δούμε δηλαδή ποια ήταν τα επιτυχημένα βήματα μέχρι τώρα. οποιαδήποτε μοντέλο, οποιαδήποτε πρότυπα έχουμε δει ότι έχουν επιτύχει, ότι είναι επιτυχημένα, νομίζω ότι ε, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω κυρίως όσον αφορά τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού ε, τομέα. Και νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το puzzle και εν πάση περιπτώσει να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβαίνοντας συναδέλφους καθώς επίσης και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ελπίζω ότι μετά το πέρας της εργασίας μου ε, θα συμφωνήσει και η βιομηχανία. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω ότι στις 21, 21 με 25 Ιουνίου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση η συνάντηση της ICANN. Επίσης, το Ίδρυμα, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, του Ίντερνετ, το οποίο προεδρεύω, ε, θα παραθέσει γεύμα με τους περισσότερους από τους ε, ηγέτες της ICAN. Και, ελπίζω, και νομίζω ότι και το Σεπτέμβριο, αν δεν, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι κυβερνήτες της ICAN θα συνεδριάσουν στην Λιθουανία. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αντιπροσωπεία και του Κοινοβουλίου Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένω όμως ε, μπορούμε να στείλουμε κάποιον εκπρόσωπο από την Επιτροπή μας, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας κάνω και κάποιες ανακοινώσεις. Αύριο ε, προσέξτε ότι θα πάμε ε, στη διπλανή αίθουσα αύριο το πρωί, στην 3G3 που είναι και πιο όμορφη και πιο μεγάλη αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε στις 9. Και μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ενιαίο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την ε, Ελβετία. Ελπίζω ότι θα είστε όλοι εδώ για να στηρίξετε και τον εισηγητή μας τον κύριο Τσρασκόφσκι ε, και εν πάση περιπτώσει επειδή θα αλλάξουμε αίθουσα εάν προσέξτε να μην ξεχάσετε τίποτα ακουστικά λέει ο πρόεδρος ε, κινητά τηλέφωνα απόρριτα έγγραφα ύψης της σημασίας έγγραφα οτιδήποτε χρειάζεται το πάρετε μαζί σας καλό σας βράδυ